gentlemen, we should start. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε γιατί ήδη έχουμε μια δεκάλεπτη καθυστέρηση. Δυστυχώς λίγα μέλη έχουν έρθει μέχρι στιγμής, αλλά συμπίπτουν ε, οι συνεδριάσεις των Επιτροπών ΣΟΥΡ, ε, Βιομηχανίας, ε, Περιβάλλοντος και έχουμε και τη δική μας ε, συνεδρίαση και την πολύ σημαντική έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη. Θα περάσω τώρα στα γερμανικά. Πρώτο σημείο. Είναι web stream τη συνεδρίαση και μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει από το διαδίκτυο. Ερωτώ αν συμφωνούν όλοι με την ημερήσια διάταξη και βλέπω ότι συμφωνούν. Άρα λοιπόν προχωρούμε στο σημείο 2 και ρωτώ για τα πρακτικά της ε, περασμένης συνεδρίασης. Εάν συμφωνείτε, αν υπάρχουν προσθήκες στα πρακτικά, προτάσεις άλλες, βλέπω όχι. Καλωσορίζω στο σημείο αυτό μια ομάδα επισκεπτών και δημάρχων από την Ελλάδα, προσκεκλημένη του συναδέλφου κυρίου Σταυρακάκη, ε, θα μου επιτρέψει να τον αποκαλέσω Γιώργο. Καλώς ήρθατε, ένα θερμό καλωσόρισμα στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή. Επειδή η πρόεδρος η κυρία Χούμπνερ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, ε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, το τυπικό καλωσόρισμα και το επίσημο θα γίνει αργότερα από την ίδια. Και περνάμε στην έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη που είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό γιατί αφορά το, τις συνέργειες ε, μεταξύ των ταμείων και του ε, Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων. Με, μεγάλη, ε, με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω τι θα μας πει ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσεκλημένοι μας, η κύρια παραδοχή που αναπτύσσεται στο σχέδιο έκθεση υποστηρίζει ότι η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη και των άλλων ταμείων θα συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην ενίσχυση τη αποτελεσματικότητα όσο και τη προστιθέμενη αξία τη πολιτική συνοχή. Ταυτόχρονα ζητείται η περαιτέρω ενίσχυση των συνεργειών με τι αναπτυξιακέ δράσει του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτική Ανάπτυξη και του Ταμείου Αλίας ενίσχυση των συνεργειών στην πράξη σημαίνει ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διάφορα ταμεία της πολιτικής συνοχής προετοιμάζονται, σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου κοινού σχεδιασμού, έτσι ώστε κάθε δράση να αξιοποιεί και να συμπληρώνει τα θετικά αποτελέσματα των άλλων δράσεων. Ταυτόχρονα, με μια τέτοια προσέγγιση αποφεύγεται η παράλληλη χρηματοδότηση μιας δράσης από διάφορα ταμεία, διασφαλίζεται το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και ενισχύεται κυρίως η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το κύριο αίτημα που διατυπώνεται στην έκθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η υιοθέτηση κοινών κανόνων διαχείρισης και εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη, το Ταμείο συνοχή και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο γενικό πλαίσιο τη πολιτική συνοχή, καθώ και με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλλία. Οι κοινοί κανόνε που θα ισχύσουν περαιτέρω στι προσπάθειε απλοποίηση, θα μειώσουν τα ποσοστά λαθών, θα κάνουν ευκολότερη τη διαχείριση και την πρόσβαση σε προγράμματα για του μικρού τοπικού φορεί, ενισχύοντας έτσι και την απορρόφηση των πόρων. Αγαπητοί συνάδελφοι, λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν θα ήθελα να σταθώ περισσότερο σε λεπτομέρειες του σχεδίου έκθεση, το οποίο εξάλλου όλοι έχετε στα χέρια σα. Πιο επικοδομητικό θα ήταν να ακούσω τα σχόλιά σας επί των θέσεων που διατυπώνονται στην έκθεση. Κλείνοντα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά σε περίπτωση υποβολής τροπολογιών να λάβετε υπόψη ότι μιλάμε για συνέργειες και μόνο ώστε να αποφύγουμε τη διατύπωση γενικών προτάσεων για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Κάτι που είχα την τάση να κάνω κι εγώ κατά τη σύνταξη της έκθεσης αυτής. Αλλά όπως όλοι γνωρίζετε, για αυτό το θέμα προβλέπεται μια ειδική έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Ο κύριος Κύριλοφ ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Σταυρακάκη για την εξαιρετική του εργασία επί του σημαντικού αυτού θέματος βελτίωσης των συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό είναι κάτι που πολύ συχνά μας απασχολεί. Εντοπίζονται από τον εισηγητή πολύ σημαντικά καυτά θέματα που αφορούν το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Συμφωνούμε ότι ο στόχος της πολιτικής συνοχής είναι να στηρίξει τα κράτη-μέλη και τις περιφερειές τους. Όμως βλέπουμε ότι πολλές φορές οι δικαιούχοι μπερδεύονται και γιατί είναι δύσκολο να γίνει σωστή χρήση των κονδυλίων των ταμείων. Επειδή υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες, προαπαιτούμενα, διαδικασίες, όταν υπάρχουν ε, διάφορα μέσα που στοχεύουν στους ίδιους ή παρόμοιους στόχους, τότε χρειάζεται καλύτερο συντονισμός και συνοχή. Πρέπει να απλουστευθούν ε, τα προαπαιτούμενα και τα μέσα. Συμφωνώ με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις στην έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη. Το κείμενο αυτό ε, γεφυρώνει τις ε, θέσεις της Επιτροπής για διάφορα θέματα που εντάσσονται στην περίοδο προγραμματισμού την τρέχουσα. Θα πρέπει τα μέσα να διατεθούν και να είναι και αξιοποιήσιμα και ελκυστικά για τους δικαιούχους. Πρέπει λοιπόν να ενσωματωθούν με βάση ένα κοινό νομοθετικό και στρατηγικό πλαίσιο. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε τους κανόνες, να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους κοινού κανόνες και χαρακτηριστικά για την τρέχουσα και επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό δεν είναι μόνο ανάγκη που απορρέει από την παρούσα εμπειρία, αλλά είναι και ανάγκη για να επιτύχουμε την, ε, τους κοινού στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, που είναι πολύ σημαντικό ε, και συζητείται αυτή την περίοδο. Υπάρχει και ένα ζήτημα βέβαια που πρέπει ίσως να το εξετάσουμε περισσότερο γιατί έχει να κάνει με την εισαγωγή νέων ε, μέσων οικονομικού σχεδιασμού, δημοσιονομικού σχεδιασμού. Ακόμα η αποτελεσματικότητά τους δεν μπορεί επαρκώς να μετρηθεί γιατί βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο υλοποίηση στα κράτη-μέλη. Ε, οι στόχοι είναι διαμφισβήτητοι, θα πρέπει όμως να δούμε τη θεσμική ικανότητα που υπάρχει κάθε φορά και η οποία μπορεί να οδηγεί σε καθυστερήσεις και αυτό είναι πολύ λυπηρό για τους δικαιούχους και για όλους. Κάθε νέα πρόταση λοιπόν θα πρέπει να στηρίζεται σε μια πολύ προσεκτική αξιολόγηση και εμπειρία όπως αποκομίζεται από την τωρινή περίοδο. Ε, ως προς αυτό θα καταθέσω ίσως μια τροπολογία. Θα ήθελα να επανέλθω στο τέλος σε αυτά που είπα στην αρχή. Είναι εξαιρετική η έκθεση, είναι πραγματικά σοβαρή συμβολή και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα δαπανίσει τον δέοντα χρόνο στην εξέταση της έκθεσης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ταξέρα. Ευχαριστώ κύριε Κύριλοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι η έκθεση που εξετάζουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όχι μόνο γιατί κάνει έναν απολογισμό της μέχρι τώρα κατάστασης των διαφορετικών ταμείων και του αναπτυξιακού ταμείου, αλλά πρώτα απ' όλα γιατί αναφέρεται στις μελλοντικές ε, συνέργειες και την ε, βέλτιστη αποτελεσματικότητα στη χρήση των ε, ταμείων αυτών. Οπότε η έκθεση αυτή και λόγω του περιεχομένου και του αντικειμένου του, αλλά και λόγω της σκοπιμότητας και της, ε, τους, της ιδανικής στιγμής στην οποία υποβάλλεται, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι συνεχίζεται η συζήτηση για τις δημοσιονομικές πρακτικές μετά το 2013, γι' αυτό και το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και λόγω της χρονικής στιγμής ε, στην οποία υποβάλλεται η έκθεση γιατί η συγκυρία είναι πολύ σπουδαία. Η έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη μας δίνει την ευκαιρία να υποβάλουμε προτάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των συνεργειών και της αποτελεσματικότητας των μέσων χρηματοδότησης πολιτικής συνοχής και υπό αυτή τη σκοπιά και υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξετάσουμε την έκθεση. Ήθελα να συγχαρώ θερμά τον κύριο Σταυρακάκη για την εξαιρετική του έκθεση και θα ήθελα να το συγχαρώ επίσης ε, για την προσήλωσή του και την επιμέλεια του ε, και την πολύ ενδιαφέρουσα εργασία του για την έκθεση αυτή και ως και όδης θα ήθελα να υποβάλω κάποιες προτάσεις προς τον εισηγητή προσπαθώντας να εμπλουτίσω κι εγώ αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι υπέρ του ενιαίου στρατηγικού πλαισίου και του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Άλλωστε αυτή είναι μια πρόταση που περιλαμβάνεται και σε μια επιστολή που είχαν στείλει επίτροποι περιφερειακής πολιτικής αλληλείας, απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και γεωργίας προς τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να βρούμε καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης μέσω κάποιων ε, χρηματοδοτικών ε, μηχανισμών και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάποιες αναλλακτικές λύσεις και το αποτέλεσμά τους εν μέσω της κρίσης στην οποία βρισκόμαστε. Επίσης γίνονται κάποιες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε την πρόταση για ένα πλαίσιο συνοχής για το ΦΕΠ και το ΦΕΝΤΕΡ, δηλαδή για το Ταμείο Γεωργίας, Περιφερειακής ανάπτυξη και Ελίες. Είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιε συνέργειες, γιατί πραγματικά στι περιφέρειες είναι που αξιοποιούνται και χρησιμοποιούνται αυτά τα ταμεία. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε και πάλι το θέμα της ε, χρηματοδότησης. Είναι πολύ επίκαιρη αυτή τη στιγμή και η έκκληση για περισσότερες συνέργειες μεταξύ των ταμείων ανταποκρίνεται και σε το αίτημα για μεγαλύτερη συμμετοχή και ανάμειξη των διαφερομένων. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε η καλύτερη διακυβέρνηση με βάση αυτό το πνεύμα συνεργασίας και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε περισσότερες συνέργειες και εμείς θα ήθελα να υποβάλω και εγώ κάποιες τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Επίσης θα πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τη σχέση της με την ε, πολιτική της συνοχής. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο εργασία του κυρίου Σαλβαδόρ Γκαρίγκα στα πλαίσια της Ειδικής Επιτροπής ε, ΣΟΥΡ για τους ε, δημοσιονομικούς πόρους μετά το 2013 και αυτό το έγγραφο εργασίας είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί λέει ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούμε προς τα κράτη-μέλη. Προσπαθώντας να δείξουμε ότι οι ευρωπαϊκές δαπάνες δεν κάνουν μια ανακατανομή των ε, κονδύλιων των ταμείων, αλλά έχουν να κάνουν με την επένδυση σε μια ανταγωνιστική και ισχυρή Ευρώπη. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφέρουμε τη σημασία τη συγχρηματοδότηση και τη ανάγκη απλούστευση των διαφόρων κανόνων. Επίση, σκόπιμο είναι να αναφερθούμε και στην αρχή τη επικουρικότητα γιατί και αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση της συνέργειας και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Θα ήθελα επίσης να έχουμε μια μεγαλύτερη εμβάθυνση τη σχέση μεταξύ των ταμείων και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, χρηματοδοτώντας κάποια πιλωτικά προγράμματα και επίσης ε, στα πλαίσια του ενιαίου στρατηγικού πλαισίου να έχουμε και ερητή μία της ανάγκης ε, να εφαρμοστεί αυτό από την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Αυτές οι προτάσεις είναι μια προσπάθεια συμπλήρωση ουσιαστικά και εμπλουτισμού της έκθεσης του εισηγητού. Οι βασικές συστάσεις του εισηγητού είναι εξαιρετικά θετικές και πολύ σημαντικές γιατί θα προβάλλουν και θα συμβάλλουν στην επιτυχία της πολιτικής συνοχής. Όπως ε, μας είπε και ο εισηγητής, θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιες ε, συνέργειες και εντός της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής ε, και τα πλαίσια αυτού του πνεύματο συνεργασία θα συμβάλλουμε και εμείς στην ενίσχυση αποτελεσματικότητα και των δικών μας εργασιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να συντομεύομαι διότι θα ε, έρθει στην ώρα του Επίτροπος ε, ο κύριος ε, Αγκουράκης είναι ο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ όσο γίνεται πιο σύντομα όλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς η παράκληση για το χρόνο καλά είναι να είναι από την αρχή ώστε όλοι να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και να μιλάμε όλοι τον ίδιο χρόνο. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Ε, όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη, ε, θα ήθελα να εκφράσω την ε, μεγάλη ανησυχία μου για το γεγονός ότι οι πολιτικές αυτές, αυτό που ονομάστηκε πολιτική συνοχής, θα συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο όπως είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και να το εκτιμήσω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος να συζητάμε αυτή την έκθεση τη στιγμή που ακόμα δεν έχει καταλήξει η συζήτησή μας γύρω από τα συμπεράσματα ε, της πέμπτης έκθεσης πολιτικής συνοχής δεν έχουμε καταλήξει συμπέρασμα, ούτε η Επιτροπή μα ούτε το Ευρωκοινοβούλιο, κατά συνέπεια μάλλον πρόωρη είναι όλη αυτή η συζήτηση. Βέβαια εγώ καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο έρχεται αυτή η έκθεση και έχω δύο βασικέ ενστάσει. πέρα από τη γενική ένσταση που έχουμε με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιεθνικών στον τομέα αυτό. Η πρώτη και βασική μου ένσταση, κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με το σημείο 4 της έκθεσης του συναδέλφου κ. Σταυρακάκη, όπου γίνεται λόγος για καλύτερη γεράρχηση των προτεραιοτήτων και θεματική συγκέντρωση των κοινοτικών και εθνικών πόρων. Αυτή η διατύπωση είναι τόσο γενικόλογη που δεν λέει τίποτα ή λέει και πάρα πολλά όσον αφορά τη δυνατότητα να γίνουν περικοπές στο όνομα το ότι δεν είναι καλή η συγκεντροποίηση και δεν είναι σαφής η στόχη. Και ένα δεύτερο ζήτημα που με ανησυχεί πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε είναι το σημείο της αιτιολογικής έκθεσης στο οποίο γίνεται λόγος ότι ήδη η Ευρώπη, η Ευρώπη έχει σέλθει από την οικονομική κρίση, δεν έχω αυτή την άποψη, και κυρίως η αναφορά στην οποία γίνεται λόγος για το ότι θα χρειαστεί να υπάρχει νοικοκύρεμα στους δημοσιονομικούς λογαριασμούς, μια δημοσιονομική νοικοκύρευση. Εάν αυτή η διατύπωση τη συνδυάσω με ε, την προοπτική να, υπάρχουν, ε, τη, να υπάρχει τιμωρία για τις χώρες οι οποίες δεν τηρούν τους όρους του Σύμφωνου ε, Σταθερότητας και του Σύμφωνου Ανάπτυξης, τότε είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όλη η συζήτηση είναι στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση. Ε, νομίζω ότι έχει ε, έρθει ο Σον Κέλλη. Ναι, κρυμμένος εδώ. Είπατε σύντομη, σύντομο θα είμαι. Θέλω να ευχαριστήσω για την πολύ καλή δουλειά των εισηγητή. Ιδιαίτερα λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και την στρατηγική 2020. Στα σημεία 10 και 11 αναφέρεται στην ανάγκη της απλούστευσης, απλοποίησης και αυτό είναι κέριο θέμα στη στρατηγική 2020. Ε, θα πρέπει να ε, υπάρξει βελτίωση 25%. Ο συντονισμός επίσης θα πρέπει να γίνει σε, όλους, σε όλες τις πολιτικές. Και θα πρέπει να γίνονται όλα σωστά, να υπάρχουν συνέργειες, ε, να ε, παρακολουθεί την νομισματική πολιτική μέσα από εκθέσεις και πάνω απ' όλα να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα, διότι αυτό είναι το σημαντικότερο που θα πρέπει να παρακολουθείτε μέσα από τους ε, μηχανισμούς. Ο εισηγητής το θέλει αυτό, αυτό επιδιώκει γιατί και εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 2020 και όλων των προσπαθειών και για να επιτύχουν οι προσπάθειες που κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Λάμπερτ Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτά που είπε ο κύριος Τεϊσέρα. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός. Στις τελευταίες παραγράφους της έκθεσής σας μιλούμε για ένα είδος συγκέντρωση των διαφόρων ροών επιδοτήσεων. Είναι αρκετά επαναστατική αυτή η πρόταση. που μιλάει για ένα είδος αναστολής αυτών των διαφόρων επιδοτήσεων. Επίσης λέμε ότι από το 2013 και μετά θα πρέπει να γίνει μια εις βάθος ε, ε, αναθεώρηση και πρόγραμμα αναπεριοχή από τα διάφορα ταμεία. Τώρα για το δεύτερο πυλώνα στην περιφερειακή πολιτική έχουμε ένα είδος ξεχωριστής γραφειοκρατίας σε πάρα πολλές περιφέρειες και έχουμε ιδιαίτερες υπηρεσίες ε, με ε, κανόνες συγχρηματοδότησης και με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικά γιατί στα πλαίσια της ε, ε, συνοχής, της εδαφικής συνοχής, το περιφερειακό επίπεδο θα είναι ένα σημαντικό επίπεδο διαχείρισης της πολιτικής συνοχής. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και εκεί σημειώθηκε ένα πολύ σημαντικό βήμα γιατί εκεί αναφέρθηκε ότι καλό θα ήταν να έχουμε προγράμματα που να χρηματοδοτούνται από πολλά διαρθρωτικά ταμεία ταυτόχρονα. Μία πρόταση θα μπορούσε, μία αντίστοιχη πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνεται και στην έκθεση, να την αναδείξουμε περαιτέρω. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση και θα ήθελα να σας παραπέμψω στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας. Κυρίες και κύριοι, και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή που συνόψισε όλες τις προτάσεις και χαιρετίζω το γεγονός ότι τονίζει την περισσότερη ανάγκη για ευελιξία και συντονισμό μεταξύ των ταμείων όπως και μεταξύ δραστηριοτήτων στα πλαίσια των διευρωπαϊκών δικτύων και το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε κοινού κανόνες για τη διαχείριση των ταμείων. Ακόμα υπάρχουν ε, ε, ανισορροπίες και δυσαναλογίες μεταξύ ας πούμε της χρήσης του γεωργικού ταμείου και άλλων. Συμφωνώ με τον κύριο Βανίστελ Ρόι, ο οποίος κατέδειξε ένα πρόβλημα στο σημείο 14 και το θέμα της οριζόντιας χρηματοδότησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να τεθούν σαφέστατα οι κανόνες Αναφέρονται κάποια εμπόδια εδώ. Δεν γνωρίζω όμως γιατί ποσοστά και γιατί μεγέθη μιλάμε. Και τέλος ε, για τις ε, εταιρικές σχέσεις νομίζω ότι όταν ζητούμε την υποβολή προτάσεων και τα προγράμματα τα ίδια θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, ποιος θα είναι ο τελικός δικαιούχος και τι δυνατότητα έχει να διαχειριστεί σωστά τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ε, και ο Γιώργος για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, μία πρόταση θα ήθελα να αναφέρω μόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους τόσο για τα καλά σας λόγια όσο και για τα επικοδομητικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη συζήτηση στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης και η μόνη απόφαση που καλούμε να λάβουμε σήμερα είναι να συμφωνήσουμε για το χρονοδιάγραμμα και τη διορία για τις τροπολογίες. Προτείνω να ορίσουμε προθεσμία για τις τροπολογίες ε, στις 3η Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Ελάχιστο χρόνο έχουμε λοιπόν, πολύ σύντομη διορία για τις τροπολογίες για να προλάβουμε εγκαίρως να ψηφίσουμε. Ολοκληρώνουμε το σημείο 4 και περνάμε στο σημείο 5 που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Λάσλο Άντορ. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω εγκάρδια στην συνεδρίασή μας κύριε Πρόεδρε και χαιρόμαστε, κύριε Επίτροπε και χαιρόμαστε που ήρθατε για να μας κοινοποιήσετε τις ιδέες σας, τις προτάσεις, το όραμά σας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και θα ήθελα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να σας δώσω το λόγο κύριε Άντορ για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, είμαι πράγματι ευγνώμων για την πρόσκλησή σας και χαίρομαι που μου προσφέρετε και μου δίνετε ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας το πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την κοινωνική, την οικονομική και την εδαφική συνοχή στην μια Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κρίση. Νομίζω πως θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου ότι χρειαζόμαστε αυτή την πολιτική συνοχή. Ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που πρέπει και μια ε, πολιτική που θα αναβάνει υπόψη είναι και τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά μέσα. Γι' αυτό λοιπόν να σας πω τις δικές μου τις απόψεις επί του θέματος αυτού. Παρόλο που η οικονομική κρίση, η χειρότερη οικονομική κρίση και τα χειρότερά της δηλαδή έχουν πλέον περάσει για τα περισσότερα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της αντιμετωπίζει μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Υπάρχει καταρχήν ο κίνδυνο ότι ακόμη και αν επανέλθει η ανάπτυξη, πολλοί θα μείνουν εκτός εργασίας. Και παρά, αν θέλετε, τις προβλέψεις, η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί πάρα πολύ λίγο, ελάχιστο δηλαδή κατά τα επόμενα χρόνια. Η πρόληψη δηλαδή αυτή τη αναντιστοιχία δηλαδή, μεταξύ των ζητουμένων και των υπαρχών των αυτών προσόντων αποτελεί μια πρόκληση. Πιστεύουμε ότι οι εργασίε οι οποίε απαιτούν υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό θα αυξηθούν κατά 60 εκατομμύρια από τώρα μέχρι το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ εκείνες που ε, είναι σε θέση, θέση δηλαδή εργασίας που καταλαμβάνονται από οι εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση θα μειωθούν. Υπάρχει συνεπώς σοβαρό πρόβλημα της ε, ανεργίας των νέων που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 21% στις χώρες της Βαλτικής, στην Σλοβακία και στην Ελλάδα Φερρυπίν φτάνει το 30% ακόμη και παραπάνω και στην Ισπανία που είναι η πλέον δραματική κατάσταση υπερβαίνει το 40% αυτή τη χρονική στιγμή. Πρέπει συνεπώς να αντιμετωπίσουμε συρωματικά και το πρόβλημα της φτώχεια. Γιατί όπως θα γνωρίζετε, 80 εκατομμύρια στην Ευρώπη ζουν κάτω από το επίπεδο. Και ο κίνδυνος τη φτώχεια για τους ηλικιωμένου και τα παιδιά ήταν υψηλότερο το 2009 από ότι το 2005. Θα μπορούσα δυστυχώ να συνεχίσω με τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να λάβει υπόψη αυτές τις προκλήσεις στη στρατηγική του 2020 και την Ευρώπη του 2020 έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή ο κοινό σκοπό, να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα των πολιτικών αποφάσεων που θα ληφθεί σε εθνικό, κοινοτικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Να πω επίση κάτι σχετικά με το ρόλο των δημοσίων πόρων και των κονδυλίων. Η απαραίτητη, αν θέλετε, ενοποίηση και παγίωση των προπολογισμών δεν θα γίνει παρά πολλά χρόνια ακόμη. Πράγμα που σημαίνει θα χρειαστεί να καταλήψουμε τον ρόλο τον οποίο χρειάζεται να παίξει η δημόσια επένδυση προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για μια υφόρο ανάπτυξη, μια βιώσιμη ανάπτυξη και παράλληλα την κοινωνική συνοχή. Πιστεύουμε ότι οι προκλήσει τι οποίε περιέγραψα θα αντιμετωπιστούν χωρί την ενεργό συμμετοχή των δημοσίων πολιτικών και των δημοσίων ταμείων. Δεν νομίζω, αλλά νομίζω ότι οι δημόσιοι πόροι θα είναι πιο λίγοι και η πρόκληση που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε σήμερα να τι αξιοποιήσουμε και να τι χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Πράγμα που σημαίνει τρία πράγματα. Να δούμε τι πραγματικές, τις βασικές προκλήσεις προκειμένου να έχουμε μια ευφυή δηλαδή και περιεκτική ανάπτυξη, να στηρίξουμε εκείνους που χρειάζονται την στήριξή μας, γιατί αυτό νομίζω θα μπορούσε να προκαλέσει και τη διαφορά και να μεγιστοποιήσουμε τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο θα πανώνται τα δημόσια χρήματα. Είμαι πεπισμένος ότι αν μπορέσουμε να δείξουμε ότι η πρότασή μας πληρεί αυτούς τους τρεις όρους, και προϋποθέσεις, τότε θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική και στρατηγική συνοχή. Έχουμε κατ' επανάληψη παρουσιάσει, αν θέλετε, του προσανατολισμού που μα έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πέμπτη έκθεση συνοχή, προκειμένου να πετύχουμε αυτά τα κριτήρια και να εξασφαλίσουμε τη συνοχή με τι συμφωνηθεί σα προτεραιότητε στο πλαίσιο τη Ευρώπη για το 2020, τη συγκέντρωση, πραγματική, αν θέλετε, ρεσιμότητα, στόχευση αποτελεσμάτων, μεγαλύτερε απορροφήσεις, απλοποίηση και καινοτόμα χρηματοδότηση. Θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω όλου για την υποστήριξή μου, για την πλήρη υποστήριξή μου και τη φιλόδοξη αυτή προσέγγιση την οποία υιοθετήσατε σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Στον περιορισμένο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα τώρα να επικεντρώσω την προσοχή μου στο ρόλο που βλέπω για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα διαφορετικά ταμεία εν γέννη. Δεν θα εκπλαγείτε αν με ακούσετε να σα λέω ότι για μένα ένα πιστικό επιχείρημα ή μια ισχυρή πολιτική συνοχή μπορεί μόνο να υπάρχει αν και περιλαμβάνει, αν θέλετε, και ένα εύρο, αν θέλετε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σαν βασική πηγή χρηματοδότηση για την απασχόληση, την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Και βεβαίω και τον, και τον κοινωνικό, κοινωνική συμμετοχή. Και ω προ αυτό, η, αυτό έχει μάλλον αποδειχθεί. Με τα κονδύλια τα οποία προσθέτει στου χώρου, στου εθνικού πόρου, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Βοηθάει αν θέλετε στο να απεκλωβιστεί το κοινωνικό δυναμικό και ειδικότερα στι φτωχότερε χώρε. Και δείχνει επίση και τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι εθνικέ προτεραιότητε και πώ υλοποιούνται. Και παίζει επίση ένα σημαντικό ρόλο, διότι διαδίδει, αν θέλετε, τι καινοτόμε προσεγγίσει και βελτιώνει την γενικότερη ποιότητα τη διακυβέρνηση. Πιστεύω προσωπικώ ότι θα μπορούσε και πρέπει να πάει καλύτερα. Έχω κατ' επανάληψη πει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να πετύχει το στόχο του ω βασική συνιστόσα τη πολιτική συνοχή αλληλεπιδρώντα δηλαδή με όλα τα υπόλοιπα ταμεία και ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο και κυρίως σε αυτό. Το κοινωνικό ταμείο διαθέτει ήδη μια ισχυρή εδαφική συνοχή, ε, διάσταση. Και να σα δώσω κάποια παραδείγματα για να γίνω σαφέστερος. Πάνω από τα δύο τρίτα των επιχειρησιακών μα προγραμμάτων είναι περιφερειακή φύσεω. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων τα εθνικά προγράμματα επίσης βρίσκουν και εντοπίζουν συγκεκριμένα θέλετε περιφερειακά τμήματα και στις οποίες συμμετέχουν και εταιρικέ σχέσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Αυστρία, Φερρυπίν, Γαλλία κτλ. Από το 1997 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τακτικά στήριξε την προώθηση της τοπικής προσέγγισης σε ζητήματα, αν θέλετε, κοινωνικού, αν θέλετε, και συμμετοχής, όπως επίσης και συμμετοχής στην αγορά εργασίας, και πρόθεση αν θέλει σύμφωνα Φερρυπίν για την απασχόληση όπως επίσης και τις ανάλογες πρωτοβουλίες. Στην τρέχουσα περίοδο το Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί δράσεις που προωθούν τις τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης και τέτοιου τους σύμφωνα σε διεθνικό, εθνικό αλλά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ έχουν τεθεί κατά μέρο για την προώθηση τέτοιου εταιρικών σχέσεων και συμφώνων πολύ συχνά σε τοπικό, αν θέλετε, και περιφερειακό επίπεδο. Συμφωνώ με την άποψη η οποία εκφράστηκε από την Επιτροπή σα ότι μία από τι προποθέσει, ένα από του όρου για την περαιτέρω ενδυνάμωση του δυναμικού και τη δυναμικότητα του κοινωνικού ταμείου είναι η βελτίωση του συντονισμού με άλλα ταμεία. Στηρίζω την ιδέα τη δημιουργία ενό κοινού στρατηγικού πλαισίου που θα μεταφράζει δηλαδή του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε επενδυτικέ προτεραιότητε και θα συντονίσει τα ταμεία καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω επίσης και υψηλές προσδοκίε όσον αφορά το δυναμικό και δυνατότητα του συμφώνου αυτού να ορίσει, αν θέλετε, τις επενδυτικές προτεραιότητε με σαφέστερο τρόπο. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει και την προσθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Πολιτική συνοχή και θα δημιουργήσει, αν θέλετε, και μεγαλύτερε συνέργειε μεταξύ εθνικού, κοινοτικού και τοπικού επίπεδου. Επιπλέον, η ευθυγράμμιση αν θέλετε, των στόχων, αν θέλετε, στην παρέμβαση σε κάθε ταμείο και λεπτομερεί κανόνε επιλεξιμότητα θα βοηθήσουν στην αποφυγή των επικαλύψεων μεταξύ αυτών, θα απλοποιήσουν, αν θέλετε, τη ζωή αν θέλετε, των δικαιούχων και θα θέσουν και τη βάση για την αξιοποίηση των συμπροματικότητων. Δεύτερον, η απαραίτητη ταφική διάσταση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει πάντα να βασίζεται σε μια πολιτική αποστολή, στην οποία έχουμε εμπιστευτεί. Θα πρέπει να ακολουθεί και να συγκεκριμένου στόχου, αν θέλετε, που συνδέονται αν θέλετε, με τι πολιτικέ προτεραιότητε τι οποίε έχουμε τάξει και έχουμε θέσει. Οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε είναι περίπλοκε και απαιτούν, αν θέλετε, και περίπλοκε παρεμβάσει. Γι' αυτό τον λόγο θα ήθελα να κρατήσω το πεδίο του Ευρωπαϊκού Κοινοταμείου αρκετά ευρύ, προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει την απασχόληση, την παιδεία δηλαδή και την κατάρτιση και τον κοινωνικό εγκλισμό ή την κοινωνική συμπερίληψη, αν θέλετε, με τρόπο ολοκληρωμένο. Αλλά η αποτελεσματικότητα σημαίνει και ισιώδη συγκέντρωση όσον αφορά τι βασικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη σχετικά με του στόχου τη Ευρώπη για το 2020. Θα ήθελα όλο ιδιαίτερο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να κάνει κάτι περισσότερο για την κοινωνική συμπερίληψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό όχι μόνο για την επίτευξη αν του στόχου μείωση τη φτώχεια, αλλά και για την πρόθεση τη απασχόληση και τη απασχολησιμότητά. Και ω προ αυτό, η πρόταση και οι θέσεις αν θέλετε της μεγάλης κοινότητας, θέλετε, το Ρώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Θα χρειαστεί να προωθήσουμε επιπλέον περαιτέρω απλοποίηση και απλούστευση. Ακούω πολύ συχνά προειδοποίησει ότι αν θέλουν μια διαχείριση που αυξήσει τα αποτελέσματα ή αν θέλετε όχι στο κόστο επιστροφή δηλαδή, θα μπορούσε να περιπλέξει τα πράγματα. Δεν συμφωνώ. Διαφωνώ δηλαδή. Οι πρόσφατε εμπειρίε που αποκομίσαμε με την εισαγωγή απλοποιημένων, αν θέλετε, μεθόδων επιστροφή δείχνουν ότι έχει τη δυνατότητα αυτό να απλοποιήσει και να διευκολύνει τη ζωή όλων. Θα ήθελα τέλο να στραφώ στο ζήτημα θέλετε, του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η λέξη κλειδί που μου έρχεται στο μυαλό, στο πλαίσιο αυτό, αν θέλετε, είναι η εξοπιστία. Διότι αν οι κατανομέ του προπολογισμού, δηλαδή για την πολιτική συνοχή και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεν αντιστοιχούν στου δηλωθέντε στόχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα ήταν κανεί διατεθειμένο να λάβει στα σοβαρά τι τεράστιε πολιτικέ συζητήσει που έχουμε όσον αφορά την Ευρώπη του 2020, τι ολοκληρωμένε κατευθυντήριε γραμμέ ή την πολιτική συνοχή. Αμφιβάλλω. Διότι αν πραγματικά πιστεύουμε ότι επενδύοντα στου ανθρώπινου πόρου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει τη ανεργία δηλαδή και του κοινωνικού αποκλεισμού και την επίτευξη των στόχων τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, ο μοναδικό τρόπο για να παραμείνουμε αξιόπιστοι είναι να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα σαφέ αν θέλετε, μια σαφή μάλλον κατανομή και αισιόδοξη κατανομή των πόρων του κοινωνικού ταμείου. Δεν έχω μια έτοιμη λύση για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, διότι τα τελευταία 20 χρόνια τα μειώθηκε από το 40% το 1999 σε 20% αυτή τη στιγμή. Βεβαίως αυτό επηρεάστηκε επίσης και από τη σημαντικότητα ανάγκη για δαπανηρέ επενδύσει στι υποδομέ στα νέα κράτη-μέλη, τα αποκαλούμενα νέα κράτη-μέλη. Ακόμη όμω και χωρί το Ταμείο συνοχή, το μερίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μειώθηκε σημαντικά. Η τάση αυτή ευθυγραμμίζεται και συνάδει με την ευρύτερη στήριξη που έχει εκφραστεί για την προώθηση των κοινωνικών αξιών και των ανθρωπίνων κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτώ, μπορούμε δηλαδή να διατρέξουμε και να πάρουμε τον κίνδυνο ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν τίποτα να πούν όσον αφορά τη σημαντικότητα της απασχόλησης, της παιδείας και του ε, συμπερίληψης, της κοινωνικής συμπερίληψης. Όλα αυτά θα καταλήξουν θέτω στο περιθώριο. Κυρίες και κύριοι, όπως η Επίτροπος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για τις πολιτικές τις ίδιες, σκοπεύω να φτιάξω ένα καλύτερο μέλλον και να βοηθήσω στην οικοδόμηση ενό καλύτερου μέλλοντο για του ε, συμπολίτε μα Ευρωπαίου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τι συνέργειε μεταξύ των διαφόρων μέσων και εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μα. Θα πρέπει επίση να δώσουμε και δυνατότητα στο κοινωνικό ταμείο με του πόρου, αν θέλετε, και τα εργαλεία που θα μπορέσουν να του επιτρέψουν, αν θέλετε, να συμβάλλει αποφασιστικά και καθοριστικά. Η κρίση και η αντιμετώπιση αυτή δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από τι επιχειρήσει για να απαντήσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Προσβλέπω στη συνεργασία μου με αυτή την Επιτροπή, με την Επιτροπή Απασχόληση και τον Ευρωπαϊκό Νουβούρου στο σύνολό του, για αν θέλετε, αυτό το τόσο αν θέλετε, δύσκολο έργο το οποίο έχουμε μπροστά μα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Επιτροπέ. Ναι, να χειροκροτήσουμε. Βεβαίω, πρέπει να το χειροκροτήσουμε. Και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Σουάρτερ είναι η πρώτη στον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ευχάριστο ότι μπορούμε να σας καλωσορίσουμε εδώ στην Επιτροπή και για να διαφημίσουμε και τα θέματά μας, σήμερα στις 6.30 θα ανοίξουμε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και νομίζω ότι όλοι που συνήθως εργάζονται σε άλλες επιτροπές και δεν γνωρίζουν πολύ καλά το ταμείο αυτό, θα έπρεπε να δουν την έκθεση, η οποία δείχνει ακριβώς αυτό που είπε ο Επίτροπος, ότι δηλαδή είναι ε, ένα ταμείο που δράσει τοπικό επίπεδο, το κοινωνικό ταμείο. Και θυμάμαι ότι η προηγούμενη ε, Κομισιόν έκανε προσπάθειες για να κατεβάσει το ταμείο αυτό στο τοπικό επίπεδο και το Κοινοβούλιο έπαιξε πρωτοπόρο ρόλο ως προς την τοπική του διάσταση ε, είχαν λάβει την οργάνωση ε, των πρωτοβουλειών ούτως ώστε η τοπική συνιστόσα να συμπεριληφθεί και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Η τοπική διάσταση έχει μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τίθενται εδώ απευθείας τα σημαντικά ερωτήματα. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή αφενός να αναπτύξουμε ένα κοινό πλαίσιο, να αναπτύξουμε κοινά δημοσιονομικά κριτήρια, γιατί έτσι το προσεγγίζουμε, και από την άλλη πλευρά να λάβουμε υπόψη μας την εξατομικευμένη, τοπική, ε, συγκεκριμένη διάσταση του Ταμείου. Αυτό θα με ενδιέφερε να το ρωτήσω σε εσά και στα πλαίσια της συνεργασίας σας με τον κύριο Χάν. Τώρα, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας σας αναφερθήκατε σε κάτι που οδηγεί σε παρανοήσει στο Κοινοβούλιο καμιά φορά. Λέτε περισσότερο κοινωνικό ταμείο και λέτε ότι αυτό δεν σημαίνει περισσότερα κονδύλια, χρήματα, αλλά μια μετατόπιση του κέντρου βάρους μέσα στο ταμείο. Και αναφερθήκατε σε κάποια παραδείγματα. Πώς θα λύσετε όμως συγκεκριμένα το πρόβλημα. Ο κύριος Χάν λέει ότι δεν θέλει να υπαγορεύσει τίποτε στα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει εκείνα να αποφασίζουν. Ξέρουμε επίσης ότι στο Φόρουμ συνοχή. Ε, πολλοί τόνισαν το θέμα αυτό, δηλαδή τις ανάγκες να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη ε, και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών το ζήτησαν αυτό. Πώς θα λυθεί αυτό, να υπάρχει αύξηση των παρεμβάσεων του κοινωνικού ταμείου και αντιμετώπιση των προκλήσεων μεσούσης της κρίσης και ε, επίλυση του θέματος της καταπολέμησης της ενεργείας, δημιουργίας της θέσεων εργασίας κλπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τις ε, παρατηρήσεις σας. Σπέβδω να πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να το προσεγγίσουμε ως ε, σημαντική ε, συνιστώσα, όμως θα με ενδιαφέρουν ορισμένε πρακτικές λεπτομέρειες. Αν εφαρμόζονται τα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου στις περιφέρειες, καλύπτεται μια τεράστια γκάμα ε, θεμάτων αρχίζοντας από την ε, ενσωμάτωση και επανεισαγωγή στην αγορά εργασίας παλαιών κρατών μένων σχολική εκπαίδευση που πρέπει να βελτιωθεί, κατάρτιση, ε, μέτρα για τους ε, μετανάστες εργαζομένους. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Εμένα θα με ενδιέφερε να μου πείτε ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητές σας για το ταμείο αυτό. Δηλαδή θα δώσετε περισσότερο βάρος στην επαγγελματική εκπαίδευση, την ε, ενσωμάτωση. Αυτό θα με ενδιαφέρε πολύ. Μια δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Στην πράξη, καλό θα ήταν να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση του κοινωνικού και του περιφερειακού ταμείου και των αντίστοιχων προγραμμάτων. Αν ένα πρόγραμμα προωθείται από κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου αλλά έχει και κοινωνική διάσταση, ε, Σήμερα είναι δύσκολο να υπάρξει κοινή χρηματοδότηση και οι διαδικασίες είναι πολύ δύσκολες. Τι σκοπεύετε να κάνετε σε αυτό το θέμα για την επόμενη περίοδο πρόθεσης των έργων των ταμείων. Επίσης, έχω μια άλλη ερώτηση. Αναφερθήκατε στις σημερινές δημοσιονομικές δυσκολίες και τα οικονομικά προβλήματα το, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχετε υπόψη σας ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου σε συνδυασμό με κάποια μορφή συγχρηματοδότηση ή θα παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λάμπερτ Βανίλστεροι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στην Επιτροπή μας είμαστε πολύ υπέρμαχοι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και μάλιστα με την ευρία έννοια που δίνουμε στον όρο κοινωνικό και οικονομικό. Θα πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής συνοχής στο κοινωνικό ταμείο. Δεν θα πρέπει να είναι ένας απομονωμένος πυλώνας. Στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Συντάστε μια έκθεση που υιοθετεί μια ισορροπημένη προσέγγιση. Θέλουμε μια οριζόντια προσέγγιση ώστε οι πυλώνες να έχουν ε, σχέση μεταξύ τους. Νομίζω ότι έτσι θα δημιουργήσουμε την ισχύ της Ευρώπης. Φυσικά τα κράτη-μέλη καλούνται να λάβουν κάποιες αποφάσεις και υπάρχει το θέμα της χρήσης ή μη χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Πάντως εμείς θα σας υποστηρίξουμε στις πρωτοβουλίες σας. Σε προηγούμενη συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή μας, είχαμε ήδη ασχοληθεί με το θέμα των κατευθυντηρίων γραμμών και σκεφτήκαμε να μεριμνήσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε μία ολοκληρωμένη πολιτική των περιφερειών, ώστε τα διάφορα ταμεία να μπορούν να χρηματοδοτούν ενιαία προγράμματα γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς περιορισμούς και διαφορές και διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τάχθηκε υπέρ μιας πολυταμιακής προσέγγισης. Ποια είναι η δική σας γνώμη. Νομίζω ότι με μια τέτοια προσέγγιση θα ελαφρύνουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Στα γερμανικά κρατήδια, για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα όργανα που ασχολούνται με το Κοινωνικό Ταμείο, άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με το Κοινωνικό Ταμείο, άλλες για το Περιφερειακό Ταμείο. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Εν ώψη λοιπόν της στρατηγικής για το 2020, πώς θα μπορέσουμε να άρουμε αυτούς τους φραγμούς και να ταχθούμε υπέρ μιας ενοποίησης και όχι αυτού του κατακαιρματισμού. Πολύ σωστά μιλήσατε για το πρόβλημα των Ρώμα. Και είπατε ότι είναι προσφυλές το θέμα αυτό για σας. Δυστυχώς τα κονδύλια που είχαμε για την υποστήριξη της κοινότητας αυτής δεν αξιοποιήθηκαν δεόντως. Πού οφείλεται αυτό σε προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σε περιφερειακό ή σε εθνικό επίπεδο. Ίσως για τις ενδιαφερόμενες χώρες θα μπορούσαμε να προβλέψουμε αυτή τη δυνατότητα ε, για διευκόλυνση της στέγασης κάποιων περιθωριοποιημένων ομάδων ε, ή κοινοτήτων. Γιατί κάτι τέτοιο ήδη αποφασίστηκε πέρυσι το Μάρτιο. Υπάρχει σχετική νομοθεσία, αλλά δεν είχαμε προσαρμογή κανενός προγράμματος. Τι γίνεται λοιπόν, γιατί δεν εφαρμόζεται η πολιτική. Μήπως δεν ανταποκρίνεται αυτή η πολιτική στις πραγματικές ανάγκες. Εγώ περιμένω μία έκθεση και έναν απολογισμό των, της μέχρι τώρα πολιτικής, ώστε να μην βρεθούμε μετά από τρία χρόνια να αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και να βρισκόμαστε σε διέξοδο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την αποκέντρωση για τη διαχείριση των ταμείων και αν δεν αξιοποιούνται κάποια κονδύλια να επανέρχονται σε ένα κεντρικό ταμείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λαμπέρτ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να σχολιάσει τις παρατηρήσεις των τριών ομιλητών. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Ελίζα Μπεθ Σρέντερ που αναφέρθηκε στα εγγένεια που θα γίνουν σήμερα της έκθεσης. Κάτι που δείχνει πώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αφορά τους ανθρώπους, αγγίζει τις ζωές των ανθρώπων και συγκεκριμένες καταστάσεις, γιατί ε, η ζωή των ανθρώπων μπορεί να αλλάξει άρδιν με μια υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από τα προγράμματά του. Και νομίζω ότι μερικά από τα παραδείγματα που έχουμε είναι πολύ συγκινητικά και πολύ χαρακτηριστικά. Φυσικά πολύ περισσότερα παραδείγματα υπάρχουν από αυτά που ε, μπορεί να δει κανείς σε μια έκθεση, αλλά και από την έκθεση αυτή βλέπει κανείς την διάσταση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην καθημερινότητα και πώς αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Κάτι που είναι πολύ πιο απτό από ότι κάποια ψυχρά νούμερα που μπορεί να ακούσει κανείς σε μια παρουσίαση. Φυσικά είναι απαραίτητο να μιλούμε και για πολιτικές και για το περιεχόμενό τους και για νούμερα. Και για μας σημείο κλειδί εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική και το 2020. Γιατί αυτή η στρατηγική θα θεσπίσει τις προτεραιότητες για το μέλλον. Στη φάση αυτή αναζητούμε τον καλύτερο τρόπο για να υλοποιήσουμε τους στόχους της στρατηγικής του 2020 και να σχεδιάσουμε την πολιτική αυτή στα διάφορα επίπεδα, το ευρωπαϊκό, το εθνικό, το περιφερειακό και θα πρέπει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων να μην εμπλέκονται μόνο οι κυβερνήσει και οι περιφέρειε, αλλά ακόμη και μη κυβερνητικέ οργανώσει. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι προφανέ, γιατί κάποια στοιχεία τη στρατηγική του 2020 και κάποιοι στόχοι του 2020 είναι αμυγό εθνικοί. Οι δικέ μου πάντω βασικέ προτεραιότητε, ε, που είναι ο πυλώνα για μια ανάπτυξη που δεν θα περιθωριοποιεί κανένα, που θα είναι συμμετοχική ανάπτυξη, είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση στην απασχόληση, στην παιδεία και να μειώσουμε την φτώχεια. Εκεί βέβαια οι περιφερειακές διαφορές είναι τεράστιες. Όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εντό τη ίδια χώρα υπάρχουν μεγάλε διαφορέ σε ό,τι αφορά τα ποσοστά απασχόληση μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Και καλό θα ήταν να έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα να εστιάσουμε τις προσπάθειες πολιτικής συνοχής γενικώ, αλλά ιδιαίτερα στο θέμα των ανθρωπίνων πόρων και τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για να υπάρχει όχι μόνο η προσφορά αλλά και η ζήτηση εργατικού δυναμικού σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία και μεγαλύτερη σπάνης πόρων. Και εκεί οι κυβερνήσεις έχουν πενιχρούς πόρους και δεν μπορούν να επενδύσουν σε συγκεκριμένες περιφέρειες για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν την πρόοδο και την ανάπτυξή τους. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν θα πρέπει να είναι ουδέτερο απέναντι στις διάφορες ε, περιφέρειες. Γιατί το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες περιφέρειες, αλλά και στις μικρότερες περιφέρειες και στις επαρχίες. Γι' αυτό και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Εγώ είμαι πέρα ε, του ισχυρότερου συντονισμού και του καλύτερου συντονισμού των ταμείων. Πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιωθούμε σε σχέση με το παρελθόν σε ό,τι αφορά αυτό το συντονισμό. Και γι' αυτό και το, κοινωνικό, ε, κοινό πλαίσιο στρατηγικής είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κοινό πλαίσιο και για μας, γιατί έτσι γνωρίζουμε τι κονδύλια προβλέπονται για τις διάφορες πολιτικές, αλλά είναι σημαντικό και για τους τελικούς χρήστες, τους δικαιούχους δηλαδή, γιατί και οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσεγγίσουν τις διάφορες δυνατότητες που τους προσφέρει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με σαφήνεια. Δηλαδή να γνωρίζουν ακριβώς τι, τι ταμείο ενδείκνεται για τον κάθε σκοπό, για το κάθε πρόγραμμα και ποια είναι η σύνθεση των διαφόρων πόρων τι μείγμα μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τους δικούς τους αναπτυξιακούς στόχους. Πρωταρχική μας προτεραιότητα είναι να υλοποιήσουμε τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από αυτά που είπα. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα γίνει κάτι τέτοιο. Πώς θα υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους του 2020. Δεν αρκεί να πούμε ότι όλες οι χώρες είναι πρόθυμες να υλοποιήσουν τη στρατηγική και τους στόχους του στόχου της στρατηγικής του 2020, γιατί οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφορες χώρες είναι ποιοτικά διαφορετικές. Κάποιες προκλήσεις για την αγορά εργασίας είναι κοινέ. Ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, το θέμα της γύραση του πληθυσμού είναι κοινό. Επίσης, αναντιστοιχία των προσόντων με τη ζήτηση. Αυτά είναι γενικά θέματα που απασχολούν όλες τις χώρες μέλη εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να μπορούμε οριζόντια να συμβάλλουμε για την βελτίωση της παιδείας, την αηφόρο κατάρτιση, για ανανεωμένε δυνατότητε επιμόρφωση και κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να παραμένει ενεργό το εργατικό δυναμικό, ιδιαίτερα σε μια εποχή που αυξάνονται οι ηλικίε ταξιοδότησης. Και χρειαζόμαστε κάποιες προσπάθειες και από την ε, πλευρά της ε, προσφοράς, αλλά θέλουμε να υποστηρίξουμε και την ζήτηση, να υπάρχει δηλαδή μια υφόρο ζήτηση για τις μειονότητες για παράδειγμα, αν υπάρχουν τεράστιες διαφορές και στα ποσοστά απασχόλησης σε μερικές ευρύτερες περιφέρειες ή μικρές περιφέρειες. Για αυτά τα θέματα λοιπόν το ΕΚΤ μπορεί να συμβάλλει με οριζόντιο τρόπο. Υπάρχουν βέβαια ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένε περιοχές ή μικροπεριφέρειες. Για παράδειγμα, αναφέρθηκα στους Ρωμά. Το πρόβλημα των Ρωμά αφορά ιδιαίτερα ορισμένες περιφέρειες ή ορισμένες χώρες. Ακόμη και αν το πρόβλημα έχει το θέμα, το ζήτημα έχει πια αναχθεί σε ευρωπαϊκό, γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά σύνορα και δεν περιορίζεται πια το πρόβλημα στη συγκεκριμένη επικράτεια εθνική. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κανονισμό που δεν θα μας επιτρέπει απλώς ένα συνδυασμό των κοινοτικών κονδυλίων, αλλά έναν συνδυασμό των κοινοτικών πόρων με άλλους πόρους. Σε άλλες περιπτώσεις είχα αναπτύξει αυτό το σημείο, θα το επαναλάβω και εδώ, γιατί πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι μια καλύτερη εστίαση, στοχοθέτηση, να κατανοήσουμε καλύτερα ε, και τους δικαιούχους αλλά και τις ανάγκες, αλλά να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τους πόρους του ΕΚΤ και με άλλες πηγές, για παράδειγμα ιδιωτικές ή με οι διεθνείς τράπεζες όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να ενισχύσουμε την χρηματοοικονομική δυνατότητα του Κοινωνικού Ταμείου και την δυνατότητα επιδίωξης των στόχων της στρατηγικής του 2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά έχει περιορισμένου πόρου και το ίδιο θα γίνει και σε επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Γι' αυτό και θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τη δική μας συνεισφορά και συμβολή με τη συνεισφορά του ιδιωτικού φορέα και των πόρων του ιδιωτικού κλάδου. Ακόμη διερευνούμε τις διάφορες αναλεκτικές λύσεις για να αναπτύξουμε αυτό το συνδυασμό, αλλά και το θέμα του δημοσιονομικού σχεδιασμού ή των χρηματοοικονομικών τεχνικών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Την περασμένη το, περισμένο Οκτώβριο μάλλον είχα πάει στο Βουκουρέστι και το πρόβλημα όντως ε, είναι σημαντικό στη Ρουμανία και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και το Αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και προσπάθησε να βρει τα εμπόδια που υπάρχουν και που παρεμποδίζουν την ε, απρόσκοπτη χρήση του ΕΚΤ. Υπάρχει όμως πρόβλημα με τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης της Ρουμανίας αλλά και με τη διοικητική ικανότητα της Ρουμανίας και κάποια προβλήματα της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να δούμε πώς θα επιλέξουμε τα καλύτερα σχέδια και προγράμματα για τη χώρα αυτή, γιατί όντως αν δεν υπάρξει επιτάχυση του ρυθμού απορρόφησης και εκταμίευσης των κονδυλίων από τη Ρουμανία, ίσως η χώρα αυτή αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να χάσει αυτά τα κονδύλια. Ναι, αλλά το θέμα είναι να μπορούν οι δικαιούχοι άμεσα να έρχονται στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν, αν δεν μπορεί η χώρα να το αντιμετωπίσει, γιατί να μην έχουμε δυνατότητα άμεση επαφή των δικαιούχων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρη αυτή η ιδέα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη ε, στη συζήτηση εναλλακτικών λύσεων με συγκεκριμένο τρόπο. Καλώς. Συνεχίζουμε με τους συντονιστέ, Ο κύριος Όλτσιχ Βλάσα και μετά η κυρία Μανέσκου. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι και εγώ που είμαστε σε θέση να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό μαζί σας σήμερα. Διότι πιστεύω ότι μία από τις προτεραιότητες είναι η αύξηση της απασχόλησης. Και πιστεύω μάλιστα ότι η χρηματοδότηση αν θέλετε, θα πρέπει να έρχεται αν θέλετε, προληπτικά και όχι να έρχεται να αντισταθμίσει. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις ανάγκες των περιφερειακών αγορών. Ταυτόχρονα όμως πρέπει νομίζω, να υπάρξουν παρεμβάσεις και από άλλα ταμεία, όπως Φερρυπίν, το Περιφερειακό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και άλλων επίσης. Πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους μικρούς επιχειρηματίες. Εσείς πάντως, τι πιστεύετε, πώς θα μπορούσαμε Φερρυπίν να συνδυάσουμε το Περιφερειακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο σε διάφορα projects τα οποία θα χρηματοδοτήσουν. Κύριε Μανέσου τώρα παρακαλώ. Να uh, uh, ευχαριστήσω και εγώ τον Επίτροπο για την παρουσίασή του, θα ήθελα. Προφανώς μιλούμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και την επερχόμενη περίοδο και αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε είναι πώς θα μπορέσουμε πιο αποτελεσματικά να τονώσουμε την ανάπτυξη, την απασχόληση και να σχηματίσουμε και να αποκτήσουμε μάλλον μια πιο βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία. Και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι αυτό του, της κοινωνικής συμπερίληψης που μάλιστα ενσωματώνεται και στις περιφερειακές πολιτικές. Και όπως έχω πει προηγουμένως, συνεπάγεται κάτι παραπάνω από η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μόνον. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει βεβαίω ένα σημαντικότερο ρόλο να παίξει προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης του 2020. Χωρίς περιφερειακά εργαλεία και μέσα, αυτή η πολιτική για την Ευρώπη του 2020 δεν θα μπορέσει ποτέ να υλοποιηθεί αποτελεσματικά, είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό, είτε και ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Ένα πράγμα είναι σαφέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα στοιχείο κλειδί ένας καθοριστικός παράγοντας στην καταπολέμηση αυτής της οικονομικής κρίσης στην οποία διέρχεται η Ευρώπη μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης βεβαίως. Και μέχρι τώρα τα δύο αυτά ταμεία συνεργάστηκαν πολύ καλά μεταξύ τους και πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον ίδιο τρόπο και ακόμη καλύτερο. Θα πρέπει, αν θέλετε, να ολοκληρωθούν με οριζόντιο τρόπο, διότι αυτό έχει ζωντική σημασία όσον αφορά το μέλλον τη πολιτική συνοχή για το μέλλον. Μιλήσατε για καλύτερο συντονισμό των ταμείων. Μιλήσατε επίσης για την ανάλυση την οποία πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον αντίκτυπο και την χρήση αυτών των ταμείων από τα διάφορα κράτη-μέλη και ειδικότερα του Κοινωνικού Ταμείου και αναφερθήκατε και στην Ρουμανία. Είπατε δηλαδή ότι στη Ρουμανία το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά τα διαστοτικά ταμεία εν γέννη τα κονδύλια του δεν απορροφήθηκαν με ικανοποιητικού ρυθμού. Είναι πολύ χαμηλό ο ρυθμός αν θέλετε απορρόφηση των κονδυλίων αυτών των ταμείων. Να ρωτήσω όμω κάτι κύριε Επίτροπε. Τι μέτρα πιστεύετε θα μπορούσαμε εμεί να λάβουμε ω Επιτροπή εδώ του Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα μέτρα δηλαδή τα οποία θα απευθύνονται στα κράτη-μέλα τα οποία αδυνατούν από διοικητική απόψεω να απορροφήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια κοινοτικά κονδύλια, γιατί κανεί δεν θέλει να τα χάσει αυτά στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Αν διαπιστώσουμε δηλαδή και δούμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που συνεχώ αντιμετωπίζουν προβλήματα με την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων, θα πρέπει να μπορέσουμε να επέμβουμε και να παρέμβουμε. Πρέπει η άμεση διαχείριση να αποτελεί, αν θέλετε, μια πιθανή λύση στο πρόβλημα αυτό. Μία από τι λύσει στο πρόβλημα αυτό, αλλά και άλλοι μηχανισμοί και άλλα εργαλεία και άλλα μέσα, τα ευρωομόλογα, Φερρυπίν, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή παράγωγα αυτών και όλα αυτά νομίζω θα μας επιτρέψουν να δώσουμε σε αυτά τα κρατημέλη να αξιοποιήσουν τα κονδύλια αυτά, να τα χρησιμοποιήσουν και να αποφύγουμε την απώλεια των κονδυλίων αυτών για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πέντε ομιλητές και 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να θέσετε τα ερωτήματά σας και μόνο. Μην μακρηγορήσετε. Λυπούμε, αλλά διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να τι θα προκάνουμε. Και θα πρέπει στις 4.30 αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Κύριε Επίτροπε, καλημέρα σας. Θα πρέπει να παρακολουθούνται τα project δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, μια πιο μακροπρόθεσμη παρακολούθηση. Γιατί αναφέρεται σε όλου του πάντε και στα ευαίσθητα άτομα και απαιτεί, αν θέλετε, μια ποιοτική προσέγγιση. Είτε μέσω της εξέλιξη, αν θέλετε, των αναγκών αθλητικά του προγράμματος επίσης και την δημιουργία των συντελεστών. Βάσει των αποτελεσμάτων τα οποία εσείς παρουσιάσατε και μας είπατε ότι η ανάπτυξη θα φροντίσει έτσι ώστε να υπάρξουν θέσεις απασχόλησης. Και λέω ότι υπάρχουν πολλές ε, χώρες μέλη στις οποίες υπάρχει ανάπτυξη αλλά βεβαίως δεν υπάρχει απασχόληση. Δεύτερον, να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν πρέπει κυρίως να εγκαταλείψει το ότι επί από κοινωνική απόψεω το ζήτημα αυτό, ότι υπάρχει ανθρώπινη διάσταση που είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη και προκειμένου να επανέλθουμε στην πλήρη απασχόληση. Η στρατηγική αυτή, όπω είπατε και εσεί, έχει σαν στόχο 20 εκατομμύρια Ευρωπαίου να του βγάλει, αν θέλετε, από τη φτώχεια στην οποία έχουν περιέλθει. Η στρατηγική Λισαβόνα, όπω είπα, θα εξαλείψει τη φτώχεια, αλλά σήμερα η έκρηξη, αν θέλετε, τη φτώχεια στην Ευρώπη αποτελεί πραγματικό γεγονό. Κύριε Επίτροπε, οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν μπορούν να αρκιστούν μόνο στι δικέ του ανακοινώσει. Ποια είναι τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα θέσει στη διάθεσή του για την εξάλληψη τη φτώχεια. Πρώτο με ερώτημα αυτό. Δεύτερον, τι θα κάνετε και πώ θα κάνετε έτσι ώστε να ασχεθεί πίεση στα κράτη-μέλη προκειμένου να θα τηρήσουν τι δεσμεύσει του. Τέλο, είπατε και βρήκα κάποια δικά σα έγγραφα, είπατε ότι η φτώχεια αποτελεί, αν θέλετε, ω σπατάλη και διασπάθηση, αν θέλετε, ανθρωπίνων πόρων. Και τώρα εδώ τι υπονοείτε, δηλαδή, ότι εκείνοι δεν είχαν θέση απασχόληση, δεν παράγουν πλούτο, άρα δηλαδή κατά πολέμηση τη φτώχεια, μόνο υπό το πρίσμα θα πρέπει να δοθεί το πρίσμα τη απασχολησιμότητα. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπε σα επισημαίνω ότι για να προωθήσουμε την πρόσβαση στην εργασία, στην απασχόληση ξεχνάτε και δεν πρέπει να ξεχάσετε την ύπαρξη αν θέλετε φτωχών εργαζομένων, συνταξιούχων φτωχών. Όλοι εκείνοι δηλαδή που βρίσκονται αν θέλετε σε αυτή την πρόσχερη αν θέλετε κατάσταση, την επισφαλή κατάσταση. Νέοι, γυναίκε. Επομένω, το πραγματικό ερώτημα είναι το εξή. Θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο ε, εφαρμογή αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να ευθύνει η φτώχεια της σε όλε τι πτυχέ και διαστάσει. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε, είπατε, τη συνέργεια μεταξύ του ΦΕΝΤΕΡ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε μια έκρηξη, αν θέλετε, των ενοικίων. Έκρηξη αυτή επίση των ε, ενεργειακών δαπανών, θέλετε, που έχουν σχέση αν θέλετε, με την ενοικίαση. Γιατί λοιπόν να μην γίνει μια ίδια προσπάθεια για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, θέλετε, ενέργειας. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, προφανώς, χωρίς την συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη περιφερειακής και όλων των μικροκυβερνητικών οργανισμών, αλλά και εκείνων, αν θέλετε, που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχεια. Διότι η στρατηγική την οποία στήσαμε υπέρ εκείνων, αν θέλετε, που στερούνται στέγης, οδηγούν, αν θέλετε, συμμετοχή γιατί όπω έλεγε ο κ. Τσενρό, οι περιστηριωμένε κοινότητε, οι Ρώμα δηλαδή, πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν. Και έχω και δύο ακόμη ερωτήματα. Πώ μπορείτε να εξασφαλίσετε, κύριε Επίτροπε, την ενεργό του συμμετοχή με τι δημοσιονομικέ περικοπέ. Πώ θα εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση όλων αυτών των ενεργειών και δράσεων και για να εξασφαλίσουμε μια οριζόντια προσέγγιση για την αποφυγή τη στόχια και για την πρόληψη αυτή, γιατί σήμερα είναι ζωτική σημασία, διότι βρισκόμαστε και κινούμαστε σε ένα πλαίσιο κρίσεω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και το γνωρίζουμε. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν να εγγυηθούμε και να διασφαλίσουμε σε όλου του Ευρωπαίου πολίτε την άμυνα δηλαδή και να προασπίσουμε αν θέλετε την δημόσια αν θέλετε υπηρεσία η οποία θα είναι σε συμφέρουσα τιμή και ειδικότερα στι απομονωμένε περιοχέ ή στι περιοχές τη Πέθρου. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, παραπάνω από τρία λεπτά δεν έχετε. Ε... Ευχαριστώ. Για να είμαι ειλικρινής, Είναι πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις της κυρίας Ντέλη που μίλησε τελευταία, αλλά δεν προλαβαίνω τόσο σύντομα να απαντήσω. Βεβαίως και εστιάζομαι και στην απασχόληση και στη μείωση της φτώχειας στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και την καταπολέμηση της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Και όταν εγκρίθηκε η στρατηγική αυτή, ε, είχαν προβλεφθεί περισσότερα μέτρα από το Κοινωνικό Ταμείο για την κοινωνική ένταξη. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προγραμμάτων έργων και δεν είναι μόνο τα δημοσιονομικά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καταπολεμήσουμε επισφαλείς θέσεις εργασίας, όπως λέτε πολύ σωστά, αλλά είναι και θέμα εργατικού δικαίου Επίσης είναι θέμα εκπαίδευσης των νέων, γιατί αυτά απασχολούν τους νέους κυρίως, που εκείνοι αντιμετωπίζουν αυτή την επισφάλεια. Για τις συντάξει έχουμε διαφορετική αναφορά, στην πράσινη βίβλο, έχουμε την πράσινη βίβλο που τη γνωρίζετε και αυτό που μπορεί να κάνει το κοινωνικό ταμείο δεν είναι να καταβάλει τις συντάξει. αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε κοινωνικές υπηρεσίες για ανθρώπους που απειλούνται από την φτώχεια συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων. Μπορούμε διάφορα πράγματα να κάνουμε για να αναπτύξουμε την ικανότητα του κοινωνικού ταμείου να, και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αναφέρατε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν λέτε ότι είναι δραματικότατη η κατάσταση, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιφέρειες που ε, βρίσκονται σε ύφεση ενώ άλλες ε, παρουσιάζουν ανάκαμψη. Γι' αυτό πρέπει να συζητούμε όχι μόνο για το κοινωνικό ταμείο, γιατί υπάρχουν κρίσιμες καταστάσεις, θα πρέπει να δούμε και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, γιατί πολλές φορές ε, ε, το Ταμείο αυτό είναι πιο σημαντικό σε ευρωπαϊκά πλαίσια για να αντιμετωπίσει την άνοδο των απολύσεων για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας και την απασχόληση, ο συντονισμός είναι θέμα κλειδί. Στην πρώτη παρέμβαση ετέθη το θέμα για τις υποδομές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα σαφές παράδειγμα γιατί θα πρέπει τα ταμεία αυτά να συντονίζονται, το κοινωνικό, το, το ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, τώρα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν και περιφερειακά σύμφωνα ανάπτυξη. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί και στα δύο ταμεία. Γιατί στις μικροπεριφέρειες όπου είναι υψηλή η ανεργία, αυτό δεν οφείλεται μόνο ε, επειδή λείπουν οι δεξιότητες, ε, εξαρτάται και το θέμα των υποδομών για να βοηθήσει την κατάσταση το θέμα της επιχειρηματικότητας που θα πρέπει να τονωθεί και πώς θα τονωθεί εάν ε, παίξει ρόλο και το Ταμείο Ανάπτυξης. Αυτό ε, δεν περιορίζεται μόνο στο ταμείο, ε, Κοινωνικό Ταμείο αλλά και το Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης. Γιατί Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές των προβλημάτων που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να επιτελέσουμε πρόοδο και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής 2020. Ε, ξαναγυρίζουμε στη Ρουμανία. Νομίζω ότι και το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα μπορούν να εντοπίσουν καλά έργα. Πολλά έργα μπορεί πολύ, πολλά πράγματα μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να βελτιώσει τη διοικητική ε, ικανότητα. Όχι μόνο στη Ρουμανία, θα ήταν άδικο να μιλήσουμε μόνο για αυτήν. Και η Βουλγαρία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει δυσκολίες σε αυτό το τομέα, όπως και άλλες περιφέρειες, όπου υπάρχει ανάγκη κάποια στήριξη για την ε, διοικητική ικανότητα. Συχνά όμω δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει επιλεγεί το σωστό έργο. Και εκεί και οι πολιτικοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορεί να ε, συμπαρασταθούν και να επικουρήσουν και ε, για το κοινωνικό αποκλεισμό. Σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να βοηθήσουμε την ανάπτυξη ε, αρχίζοντας από την παιδεία, την παρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού από το σχολικό σύστημα και από τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να το απασχολήσει το Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σαγκουράκης και μετά ο Μάρκος Πίπερ. Και παρακαλώ, ένα λεπτό ή δυνατόν, συνάδελφοι. Ναι, κυρία Πρόεδρε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Θα ήθελα ε, να θέσω δύο ερωτήματα στον κύριο Επίτροπο. Ε, το πρώτο ερώτημα είναι το εξή. Πώ εξηγεί ο κύριο Επίτροπο ότι η πλειοψηφία των θέσεων εργασία, οι οποίε ε, είχαν δημιουργηθεί στην Ελλάδα με πόρους του Κοινωνικού Ταμείου είναι επιτοπλίστων θέσεις επισφαλούς εργασίας, είναι συμβάσεις περιορισμένου χρόνου, θέσεις εργασίας χωρίς δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Αυτό λέει η εμπειρία της χώρας μου και το παράδειγμα που ε, ανάφερε για τη Ρουμανία ισχύει για την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Ρουμανία που δεν απορροφά όλα τα κονδύλια, είναι και η Ελλάδα και δεν τα απορροφά γιατί υπάρχει μια πολύ άσχημη δημοσιονομική κατάσταση η οποία είναι και αυτή η συνέπεια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη ερώτηση στον αξιότιμο κύριο ε, Επίτροπο έχει να κάνει με το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας για το οποίο ακούμε τόσα πολλά και το οποίο μάλλον θα υιοθετηθεί στις 11 του Μάρτη ή στις 25 του Μάρτη. Αυτό το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας κύριε Επίτροπο όπως γνωρίζετε βάζει ως απόλυτο κριτήριο των οικονομιών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Με αυτά τα και μια σειρά από μέτρα που θα αφορούν και την απασχόληση και τους μισθούς. Εσείς θα κάνετε κάτι να αντισταθείτε σε αυτό το αντικοινωνικό σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, διότι η εφαρμογή του θα σημαίνει εκτείναξη της ανεργία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρω πώς θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ, Μάρκους Πίπερ. vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Ακούγοντας κάποιους συναδέλφους, πραγματικά δεν σας ζηλεύω καθόλου. Η κοινωνική πολιτική, η πολιτική παιδείας ε, θα έπρεπε να έχει προσεγγιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτό νομίζω ότι θα ε, επιβάρυνε πολύ τις ε, πολιτικές μας. Άκουσα αυτά που είπατε για την στιβαρή προοικοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μιλήσατε και για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θέλω να την ε, εξειδικεύσουμε λιγάκι. Είμαι και εισηγητής για το πέμπτο πρόγραμμα τι σημαίνει προστιθέμενη αξία όταν μιλάμε για θέματα υγείας, ανάπτυξης των πόλεων, των μειονοτήτων, των αστέγων, ε, των ε, παιδιών που διακόπτουν το σχολείο. Και τώρα τα, το, τα διαθέσιμα ευρώ κατέτος είναι 10-20 ευρώ. Και πρέπει να καλύψουμε όλα αυτά τα θέματα. Πού βρίσκεται λοιπόν η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πού βρίσκεται ο μοχλός ο οποίος θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τα ελάχιστα αυτά κονδύλια που ελπίζω να παραμείνουν. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια προστιθέμενη αξία από τα χρήματα αυτά τα οποία δεν θα πρέπει να κατασπαταληθούν αλλά να δώσουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Σον Κέλλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον, Επίτροπο καταρχήν για την ενδιαφέρουσα σημερινή παρουσίαση που είναι και πολύ λογική. Χάρηκα που άκουσα να αναφέρει τη διαχείριση που θα στηρίζεται στα συμπεράσματα, γιατί συνάδει και με αυτά που έλεγε ο κύριος Σταυρακάκης για την απλοποίηση στην εφαρμογή και τη χρήση και τη διαχείριση των ταμείων. Ελπίζομαι ότι όλα αυτά θα τα καταφέρουμε, γιατί αφορούν τη στρατηγική 2020. Μια ερώτηση. Με ενδιαφέρον άκουσα αυτά που είπατε για τη φτώχεια αν τον ερμηνεύω σωστά, είπε ότι τώρα είναι πολύ περισσότεροι οι φτωχοί, αυτοί που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας από ότι το 2005. Για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου εδώ. Πώς μπορούμε, αν ισχύει αυτό, πώς μπορούμε να το παρουσιάσουμε αυτό στην κοινή γνώμη και ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να ε, καταπολεμήσουμε με πολλά κονδύλια την ε, φτώχεια. Δηλαδή ε, η φτώχεια παρόλα αυτά από τον τρίτο κόσμο εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, μίλησε για την κοινωνική ένταξη, για ενσωμάτωση. Ίσως ο γνήσιος αθλητισμός είναι το καλύτερο μέσο για να επιτευχθεί αυτό και εδώ αναφέρομαι και στην ε, Ιρλανδία από όπου, όπου ισχύει αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε λοιπόν ε, στα διάφορα έργα τον αθλητισμό για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα την προσπάθεια κοινωνικής ένταξης. Ο κύριος ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, όλοι επιζητούμε αποτελέσματα και είναι αναφιβολό ότι η περιφερειακή διάσταση, η τοπική διάσταση και ιδιαίτερα η ελαστικότητα και η δημιουργικότητα είναι ο καλύτερος τρόπος για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων. Εγώ κατάγομαι από μία ε, εξόχως από απόκεντρη περιοχή που έχει 6,7% ε, ανεργία. Γιατί ε, χάρη στην τοπική διάσταση μπορούμε να εστιαστούμε καλύτερα μέσω των δημοσκοπήσεων και των απογραφών στις, στις ανάγκες, στις, στη ζήτηση. Κάνουμε καλύτερο σχεδιασμό και επαγγελματικό προσανατολισμό και χάρη στην τοπική αυτή και περιφερειακή διάσταση διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερα τα προβλήματα και καταφέρουμε και αποτελέσματα σε πολιτική, στην πολιτική της απασχόλησης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Βέβαια, το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας θα είναι πιο εύκολο να το διαχειριστούμε από το Ταμείο Σταθερότητας ή Λιτότητας. Περιμένουμε πολλά πάντως από το Κοινωνικό Ταμείο για την επιδίωξη αποτελεσμάτων. Ο Αλέν Καντέκ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο τελευταίος ομιλητής στον κατάλογο. Όχι, όχι, δεν ήθελε καν το λόγο ο κύριος Καντέκ. Ο κύριος Επίτροπος, σας ευχαριστώ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πάω στην Ελλάδα, οπότε και θα έχω την ευκαιρία και η διεισόμαση να διαπιστώσω τι λειτουργεί σωστά και τι πάει στραβά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πάντως, ε, μερικά από τα σχόλια του κυρίου Αγκουράκι, δεν είναι κατά ανάγκη ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, ούτε ίδια της Ελλάδας. Το πρόβλημα ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο παρελθόν ότι δεν είχε βιώσιμα αποτελέσματα ή φόρα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν υπήρχαν ορατά και μόνιμα αποτελέσματα στο παρελθόν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις γιατί υπάρχουν προβλήματα ε, υπό αυτό το πρίσμα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό ήταν και βασικό σημείο. Μία πιθανή απάντηση είναι να χρησιμοποιήσουμε την επιμόρφωση, τη διαβίου κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση περισσότερο. Φυσικά αυτή είναι μία πτυχή της αντιμετώπισης του προβλήματος. Θα πρέπει να εξετάσουμε και το πρόβλημα σε διάφορες περιφέρειες και να δούμε ποιες είναι πραγματικά οι πηγές του προβλήματος. Αλλά θα μεταβώ, όπως σας είπα, στην Ελλάδα αργότερα μας τη βδομάδα, γιατί νομίζω ότι το καλύτερο είναι να διαπιστώνουμε την κατάσταση επιτόπου και η Κύριε Άλβες, το Δεκέμβρη είχα πάει στην Πορτογαλία και συμφωνώ ότι τα περισσότερα προγράμματα καλύτερα τα αναπτύσσονται και τα διαχειρίζονται οι περιφέρειες σε τοπικό επίπεδο. Γιατί οι ντόπιοι είναι που γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα και άρα και τις λύσεις. Και μάλιστα η Πορτογαλία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και υποδειγματικό παράδειγμα ότι το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να θεωρηθεί σε ευρύτερο πλαίσιο. Και νομίζω ότι η Πορτογαλική κυβέρνηση χρησιμοποίησε πολύ σωστά τα, τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου για διάφορα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή ένταξης ε, στην αγορά εργασίας ε, των αναπήρων, για παράδειγμα, οι άνθρωποι με ανάγκες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφήσουμε τη διακριτική ευχαίρεια και στην κυβέρνηση να παίξει το ρόλο της, σχεδιάζοντας το καλύτερο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα βέλτιστα προγράμματα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχή. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθερότητα, το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, συγγνώμη, που ήταν και μια ερώτηση του κ. Αγκουράκη. Εγώ λέω να περιμένουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μετά να επανέλθουμε στη συζήτηση ε, της γάλλο-γερμανικής, όπως τη λέμε, πρότασης. Και με το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας Είπα, είδαμε και κάποια στοιχεία που εμφανίζονταν και στις προτάσεις για, τις, ε, για την οικονομική διακυβέρνηση, για την Ευρώπη του 2020, αλλά στο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας ε, υπήρξε ένα συμπίλημα περισσότερο αυτών των μεμονωμένων ε, προτάσεων που είχαμε δει και σε άλλες προηγούμενες περιπτώσεις. Το θέμα των συντάξεων, που είναι κάτι πιο κοντά στι αρμοδιότητέ μου, νομίζω ότι εκεί έχει γίνει πολύ πιο εξεζητημένο και κλειτισμένο έργο σε θέματα συντάξεων και το συζητήσαμε αυτό και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να το αναγνωρίσουν αυτό οι συντάκτες του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας. Να αναγνωρίσουν την ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά βλέποντας και κάνοντας. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες πώς μέσω μιας συλλογική προσπάθειας θα δούμε για τις λεπτομέρειες αυτής της πρότασης. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για ένα πιο εύρωστο και ρωμαλαίο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με ευρύτερε αρμοδιότητες και με ευρύτερη προσέγγιση, αυτό δεν σημαίνει ότι το ΕΚΤ θα χρηματοδοτεί τους πάντες και τα πάντα σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα αναφερθεί σε κάποια εκπαιδευτικά ζητήματα όταν έχουν αυτά σχέση άμεσο δεσμό με τις προκλήσεις της στρατηγικής του 2020 και όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ της δυνατότητας χρηματοδότησης των τοπικών ή περιφερειακών αρχών και όταν υπάρχει άρρηκτος σύνδεσμος με άλλους στόχους, στην περίπτωση αυτή με το θέμα της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τότε στις, στα περισσότερα κρατημέλη το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Αλλά φυσικά θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε, γιατί δεν μπορούν όλες οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να υλοποιήσουν τους ε, στόχους τους, ε, να ανταποκριθούν ε, στις ανάγκες και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους χωρίς την κοινοτική υποστήριξη. Δεν σκοπεύω να μεταβώ στη Βόρεια Ιρλανδία σύντομα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο θα πάω στην Ιρλανδία, στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Βέβαια όντως αυτό είναι μια πολύ διάζουσα πρόκληση και υπάρχει ένα περίπλοκο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα και μια σημαντική πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο με το Κοινωνικό Ταμείο αλλά με ολόκληρο το οπλοστάσιο των περιφερειακών πολιτικών για να βρούμε ένα οδικό χάρτη ένταξης για παράδειγμα. Και αυτό ίσως χρειάζεται στην Βόρεια Ιρλανδία ένας μακροχρόνιος ορίζοντας όπως αυτός της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των συναδέλφων, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Θα συνεργαστούμε στενά και με εσάς και με τον Επίτροπο Χάν ιδιαίτερα στα πλαίσια της συζήτησης για τους νέους κανονισμούς και το στρατηγικό πλαίσιο. Μπορείτε να υπολογίζετε σε μας εδώ Ελπίζω ότι θα υπάρξει συνεργασία και μεταξύ των επιτρόπων που ενέχονται στις πολιτικές αυτές, γιατί για την επιτυχία χρειάζεται καλός συντονισμός και διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των επιτρόπων. Ευχαριστούμε πολύ και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στην προθυμία και τιμότητά σας να έρχεστε όποτε αυτό χρειάζεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Να δούμε καταρχήν να λειτουργούν οι κάρτες. Λοιπόν, για να χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες στο σύστημα. Ελέγχουμε αν είναι εντάξει το σύστημα. Άρχεται η ψηφοφορία. 29 κάρτες είναι στο σύστημα. Δεν ξέρω αν σημαίνει ότι είμαστε 29 μόνο σήμερα. 31 είμαστε για να ψηφίζουμε Οι πολιτικές ομάδες λοιπόν ας συντονιστούν. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. 32 ψηφίζουν. Ασυνήθιστα χαμηλό νούμερο. Για να δούμε οι πολιτικές ομάδες τι θα, ε, πώς θα ελέγξουν αυτόν τον αριθμό ε, για να ψηφίσουν όλοι όσοι δικαιούνται. Ψηφίζουμε λοιπόν έκθεση Καρόνα. Ευρώπη ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. 89 τροπολογίες υπευλήθησαν, καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές. Όμως και αρχίζουμε με τη συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προχωρούμε. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προχωρούμε στην τροπολογία 12 υπέρ κατά, αποχές δεκτή, τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 18, Α, εδώ υπάρχει μια προφορική τροπολογία «Ψηφίζομαι όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προχωρούμε. Τροπολογία 3 συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 24 υπέρ. Κατά. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε την 24 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 17 υπέρ, 14 κατά, δεκτή. Πάμε στην 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 30 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 15 προς 17. 17 κατά. Πάμε στην 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και προχωρούμε στην 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά αποχές απο, ε, δεκτή συγγνώμη 44 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω ελέγχουμε την 44 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 16 προς 15 δεκτή Προχωρούμε. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 48 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε τη 48. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16 προς 16 σημαίνει ότι απορρίπτεται, έτσι δεν είναι. Κρίμα. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 53. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 56. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τώρα ε, συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά συγγνώμη ελέγχουμε ψηφίζουμε την 66 ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία πέρας απερίφθη 16 υπέρ 17 κατά προχωρούμε 67 67 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 78 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 79 αυτά είναι γλωσσικά αφορά μόνο το αγγλικά υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται έχει πάμε στην 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ κατά Νομίζω ότι απερίφθη. Ε, ναι, απερίφθη. Να ελέγξουμε. Καλά. Αν θέλετε, ηλεκτρονική. Ε, ψηφίζουμε την 82 με ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Βέβαια, 19 είναι τα κατά, 12 η ψήφη υπέρ, απερίφθη. 83 υπέρ, κατά, αποχές, δεν ξέρω. Ψηφίζουμε την 83 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 17 προς 19. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 86 πάλι είναι μια γλωσσική για τα αγγλικά υπέρ. 86 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρουμε και παρόλο που είναι γλωσσικό το θέμα για τα αγγλικά μόνο. Τέλος πάντων ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 86. Πέρας. Δεκτή. 19 προς 15. 87 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Να δούμε. 87 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. 17 προς 15 δεκτή. Και η 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αυτή θα γίνει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 32 προς 1. Δεκτή συγχαρητήρια κύριε Καρόνα. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Ε, Όλτριτς Βλάσακ, συντάκτης γνωμοδότησης. 53 τροπολογίες αρκετές και 5 συμβιβαστικές. Και αρχίζουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές δεκτή. Δύο. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τέσσερα Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πέντε Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία επτά Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Τροπολογία 9, συγγνώμη. Τροπολογία 9, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως εγκρίθηκε. Ελέγχουμε παρακαλώ την τροπολογία 9. Ψηφίζουμε. 29-9. Εγκρίθηκε λοιπόν. Τροπολογία 10. Και υπάρχει και η μοιρασμένη ψηφοφορία εδώ. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ τώρα. Τροπολογία 13. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. 14 τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. 19. Μάλλον τροπολογία. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. 22. Τροπολογία 22. Υπέρ παρακαλώ. Τη τροπολογία 22. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγγνώμη, συγγνώμη, Νταϊάννα. Έκανα κάτι λάθος, Νταϊάννα. Τροπολογία 18. Τροπολογία 18. Τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω πως θα κάναμε τα πράγματα σωστά. Συμβαστική 3. Παρακαλώ. Για την τροπολογία παριθμών 20. Μιας γιατί ψηφίσαμε την 18. Η 16 δεν κάνει να, την 20 να, να φύγει. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ τροπολογία 20 να ψηφίσουμε. Τροπολογία 20. Ψηφίζουμε συνάδελφοι για την τροπολογία 20. Υπέρ. Της τροπολογίας 20. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ παρακαλώ. Συμβαστική 3. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Τροπολογία 42. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία 45. 46 τροπολογία. Υπέρ. 46. Κατά. Και ελέγχουμε τη 46. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας αυτής απορρίπτεται 19 προς 15. 47 η τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Τροπολογία 48. Ε, ας ελέγξουμε. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Για να κοιμάται καλά και ο κύριος Καντέξ. 48. Τροπολογία 48. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 προς 13. Έχετε δίκιο λοιπόν. 49 η τροπολογία. Μια προφορική τροπολογία. Δεν είναι κανείς κατά. Υπέρ. Κατά. Ποιο είναι κατά. Ουδή. Εγκρίνεται λοιπόν. 50. Υπέρ της 50. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα συνολικά. Έναρξη ψηφοφορίας. πέρας ψηφοφορίας δεν θα πρέπει να εκπλήσετε κανείς ότι εγκρίθηκε 33 προς 1. 33 ψήφοι υπέρ. Μία κατά. Πάμε τώρα στην επόμενη γνωμοδότηση. Αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε. Η κυρία Κονή δεν είναι εδώ. Και εδώ έχουν καταληθεί αρκετές τροπολογίες. 67 και οι συμβαστικές προτάσεις επίσης. Ξεκινάει η ψηφοφορία λοιπόν. Για την ενιαία αγορά, για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η συμβαστική τροπολογία είναι ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. is Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 16 ψήφους υπέρ, 18 κατά. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά τις 3. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 με προφορική τροπολογία. Είναι κατά της τροπολογίας κα, κανείς. Όχι. Ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ της 10. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροποποιημένη με προφορική τροπολογία 10. τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ και 12 κατά. Συμβεστική τροπολογία 3, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14, ποιος είναι υπέρ της 14, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18, ή μάλλον όχι, συμβαστική τροπολογία 4 λέει η πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον απορρίπτεται. Αν δεν επιμένει κανείς για ηλεκτρονικό έλεγχο, θεωρώ ότι απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας 2. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Ποιος είναι υπέρ. Δεν καταπίπτει. Ποιος είναι υπέρ της 37. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Ποιος είναι υπέρ Περ. ή ε, μάλλον ψηφοφορία κατά τμήματα έχουμε εδώ. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα για τη 46 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα τη 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 21 ψήφισαν υπέρ και 13 κατά εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Τι κάνουν οι σοσιαλιστές. So we parts, Επανάληψη της ψηφοφορίας για το τρίτο τμήμα της τροπολογίας 46. Παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Α, συγγνώμη, λάθος λέει πρόεδρος. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία, συμβαστική 9. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος. 33 ψήφισαν υπέρ και ένας κατά. Εγκρίνεται. Σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ελεγγύης για πλημμύρες στην Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία και Ρωμανία. Μία ψηφοφορία θα πραγματοποιήσουμε μόνο. Ποιος είναι υπέρ. Ε, ηλεκτρονικά όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Και ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Περνάμε τώρα στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, στην ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Dirk Άνερ. Ελπίζω να έχει έρθει. Σε πέντε λεπτά. Τι, τι πέντε λεπτά, δύο λεπτά, τρία λεπτά. Περιμένουμε. Εν αναμονή λοιπόν του Γενικού Διευθυντού Ας ε, ολοκληρώσω τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Σας χρωστάω δύο ανακοινώσεις. Η μία φορά την πρώτη συνεδρίαση της ε, ομάδας εργασίας για την ερεσιμότητα που έγινε στις 11 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Μια ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε μετά το Συμβούλιο του Νοεμβρίου στη Λιέγη και στην ομάδα εργασίας αυτή, εκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε η πρώτη συζήτηση το Φεβρουάριο, στις 11 Φεβρουάριο όπως σας είπα και η δεύτερη συνεδρίαση θα γίνει στις 16 Μαρτίου. Θα πρότεινα λοιπόν να σας στείλουμε ενημερωτικά σημειώματα σε όλους για το περιεχόμενο της συζήτησης. Εγώ έλαβα μέρος στην πρώτη συνεδρίαση και μάλιστα έχει προσκληθεί και η Επιτροπή απασχόληση που έδωσε το παρόν σε διοικητικό επίπεδο. Ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση. Η πλειοψηφία των κρατών μελών υποστηρίζουν αυτή την αρχή της αιρεσιμότητας. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την αρχή και όχι κατά πόσο τη χρειαζόμαστε. Ως προς την ανάγκη ήταν όλοι σύμφωνοι για τον τρόπο εφαρμογής υπήρχε συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας στέλνει σημείωμα όπως ήθιστε το δεύτερο σημείωμα θα σας το στείλουμε μόλις φτάσει. Και η δεύτερη ανακοίνωση που μας επέμεινε αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού. Οι συντονιστές, από ό,τι ξέρετε, συμφώνησαν να γίνει συζήτηση με προφορική ερώτηση και ψήφισμα στην Ολομέλεια του Μαρτίου, στο Στρασβούργο. Έχετε λάβει το σχέδιο αυτού του ψηφίσματος. Το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, μοιράστηκε. Μία τροπολογία μόνο έχουμε λάβει από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Οπότε θα πρότεινα η Επιτροπή μας να εξουσιοδοτήσει τους συντονιστές, να οριστικοποιήσουν τη μορφή του σχεδίου αυτού του ψηφίσματος και κατόπιν θα το παρουσιάσω εκ μέρους της Επιτροπής στην Ολομέλεια. Οπότε θα έχουμε και την προφορική ερώτηση με τα στο Στρασβούργο. Αν έχετε εμπιστοσύνη στους συντονιστές, μπορούμε να τους αναθέσουμε αυτό το έργο της οριστικοποίησης του ψηφίσματος μετά την τροπολογία που υπευλήθη. Αυτά με τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε ακόμη όμως το Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Dirk Άνερ.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 Uh, Κύριε Ματούλα, πως είστε έτοιμος να διεκπαιρώσουμε τη δική σας έκθεση, γιατί περιμένουμε ακόμη το Διευθυντή. Και από ό,τι ξέρω, η δική σας γνωμοδότηση είναι μάλλον σύντομη. Είστε έτοιμος τώρα να την παρουσιάσετε. Καλώς, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 14 της ημερήσης διάταξης, εν αναμονή του Γενικού Διευθυντού. Και μια και θα είναι σύντομη η παρουσίαση της γνωμοδότησης του κύριου Ματούλα, μπορούμε να το διεκπεράσουμε αμέσως. Γιώση, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως μπορώ να υποβάλω μια πολύ σύντομη παρουσίαση της γνωμοδότησης. Μια και έχουμε ε, μια πρόταση αναθεώρησης ενός πολυτεχνικού κανονισμού. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η παρουσίασή μου μπορεί να είναι λακωνική. Πρόκειται για πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προσπαθεί να θεωρήσει το κανονισμό 1698 ε, του Συμβουλίου για την υποστήριξη στήριξη αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι λογικό μετά την θέση εφαρμογή της νέας συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρειάζονται πολλές ε, τροποποιήσεις και απλουστεύσεις διαφορών κανονισμών. Με βάση λοιπόν την συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρμοδιότητες που και της ε, αρμοδιότητας τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θεσπίσει ομοιόμορφες διατάξεις για την εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, χρειάζονται κά... χρειάζεται θεώρηση του κανονισμού 1698. Επίσης, ε, θα πρέπει να πλουστευτούν κάποιοι κανόνες ε, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των προγραμμάτων και σχεδίων. Θα πρέπει να πλουστευτεί και η ΚΑΠ και οι συνοπτικές εκθέσεις να μειωθούν από 3 σε 2. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής για, τους ομάδες, για τις ομάδες παραγωγών. Δεν είναι οι τελευταίες χώρες που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ενδιαφέρονται για το σημείο αυτό, αλλά και οι 15 πρώτες χώρες, κυρίως για τα απορροκυπευτικά Επίσης ε, γίνεται κάποια απλούστευση των υπηρεσιών ε, συνδιαλλαγής. Επίσης γίνεται λόγος των ε, γραμμικών χαρακτηριστικών για το πρόγραμμα Natura 2000 προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των διατάξεων που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη στις ε, χώρες που έχουμε κάποιες ε, ειδικές ζώνες ε, προστασίας και τις επενδύσεις που χρειάζονται. Σε περίπτωση που δεν γίνεται σεβαστή αρχή της οικολογικής ρεσιμότητας θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα να δοθούν ενάβσματα με βάση το άρθρο 43 της συνθήκης που άπτεται της ενίσχυσης και των ε, όρων χορήγησής της. Κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε προβλήματα με την τεχνική αυτή, όπως σας είπα, αναθεώρηση του κανονισμού 1698, γιατί χάρη στην τροποποίηση αυτή θα έχουμε νέες βάσεις που θα συνάδουν και με την νέα συνθήκη για την εφαρμογή της Ένωσης. Γι' αυτό και κατέθεσα προς το παρόν τρεις μόνο τροπολογίες που στόχο έχουν να διευκρινίσουν τρεις τομείς δραστηριοτήτων. Εξασφαλίζουμε μια ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών μας αναγκών και των οικονομικών μας επιταγών. Ουσιαστικά οι τροπολογίες αυτές συμπληρώνουν το κείμενο και δεν το τροποποιούν άρδιν. Επίσης, τα θέματα συνδιαλλαγής στο γεωργικό τομέα. Πολλές επενδύσεις έχουν γίνει στη, στο ευρυζωνικό, στις ευρυζωνικές υπηρεσίες για το διαδίκτυο. Οπότε, θα πρέπει να προσθέσουμε και την πληροφορική εδώ και να έχουμε πραγματικά μία πύλη συνδιαλλαγής ε, για τους αγρότες μέσω του διαδικτύου για να καλύψουμε και τις εξόχως απόκεντρες γεωργικές περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις, ε, τεχνολογία, τις τεχνολογίες της πληροφορικής και να επεκτείνουμε την ευρυζωνία και στις γεωργικές ζώνες. Θα πρέπει επίσης να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των διατάξεων του Natura 2000 και των αναπτυξιακών μας αναγκών. Θέλουμε να προσφέρουμε περισσότερη ενημέρωση σε αρχικό στάδιο για την έναρξη των προγραμμάτων δηλαδή σε γεωρικές ζώνες ώστε να αποφύγουμε υπερβολικό άχθος και συμπληρωματικές δαπάνες και να αποφύγουμε και τις περιπλοκές που μπορούν να ανακύψουν στο μέλλον. Θέλουμε επίση να αποφύγουμε διαφορές και δυσαρμονία μεταξύ των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων της τοπικής και οικονομικής ανάπτυξης. Μιλήσαμε και για την χρηστή διακυβέρνηση και σε οριζόντιο και σε κατακόρυφο επίπεδο. Θέλουμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και μάλιστα σε εθνικά δίκτυα αγροτικής ανάπτυξης, η χρηστή διακυβέρνηση είναι επιτακτική ανάγκη. Σε αυτά τα εθνικά αγροτικά δίκτυα χρειαζόμαστε συμμετοχή όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και θα πρέπει η συμμετοχή αυτή να καλύπτει, όπως σας είπα, όλα αυτά τα επίπεδα. Αλλιώς δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε μια ισορροπημένη ανάπτυξη. Αυτές θα είναι συντομία οι βασικές ε, αρχές της γνωμοδότησης. Ε, Ευχαριστώ πολύ, ο Ιώσιφ, ο κύριος Αγκουράκης. Ο Σκιώδης, η Σκιώδης δεν είναι εδώ, ο κύριος Αγκουράκης. Κύριε Πρόεδρε, ε, θεωρώ ότι δεν είναι όλες οι συμπληρώσεις ε, τεχνικής φύσης, είναι και ορισμένες πολιτικές, είναι ένα άλλο θέμα τώρα πώς θα τις αξιολογήσει κανείς. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ματούλα όμως το εξή συγκεκριμένο. Η πρόταση που κάνει σχετικά με το Natura 2000 θα διευκολύνει ή θα δυσκολέψει την αγροτική δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές, θα βελτιώσει ή θα χειροτερέψει τα μέτρα προστασίας Natura 2000. Εγώ δεν κατάλαβα και θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Any other comment? Άλλα σχόλια υπάρχουν. Παρακαλώ. Η κυρία Ντελή. Euh, Απλώς για να θυμίσω κάτι το οποίο έχει τη σημασία του προς τον κύριο Συγητή. Για την τροπολογία υπάρχουν δύο θα μπορούσατε να μας διασφαλίσετε και να μας εγγυηθείτε ότι μια νέα σύνταξη, μια νέα διατύπωση θα μας επιτρέψει το περιβάλλον να μην αποτελέσει το πτωχό συγγενή αυτής της τροπολογίας, παρακαλώ. Uh, thank you. Joseph, like to, to Ευχαριστώ. Ιώσιπ, θα απαντήσεις. Η μόνη απόφαση που θα λάβουμε αφορά την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Έχετε το υπόψη σας. Υπάρχει χρόνος για κατάθεση τροπολογιών. Όσοι υπέχει το λόγο. Γιώσιφ. Ευχαριστώ. Είναι ευπρόσδεκτες οι ερωτήσεις. Μπορώ να απαντήσω. Τώρα για τις τροπολογίες που πρότεινα αναφέρεται και καλύπτεται το θέμα Natura 2000. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει λοιπόν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ των διατάξεων που αφορούν το περιβάλλον και τις τοπικές αναπτυξιακές ανάγκες. διευκρινίζω ευθύς εξ αρχής ορισμένα έργα για τα ευρωπαϊκού επίπεδου έργα. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, το τονίζω αυτό. Και αυτό στην αρχή κάποιων έργων. Αυτό περιέπλεξε και τα ίδια τα έργα. Εδώ η τροπολογία λέει μόνο ότι θα πρέπει να δώσουμε πρόσθετες πληροφορίες ώστε να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο των επενδύσεων ε, δεν θα επηρεαστεί από περιβαλλοντικές διατάξεις που υπάρχουν αλλά που δεν τις ήξεραν οι ενδιαφερόμενοι. Δεύτερη ερώτηση. Δεν πιστεύω ότι είναι φτωχό συγγενής εδώ το περιβάλλον. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα ζημιώσει από αυτή την τροπολογία το περιβάλλον. Ορίστε κυρία Ντέλη. Όταν διαβάσω την τροπολογία υπαριθμών 2 και τη λέει η τροπολογία υπαριθμών 2, υπογραμμίζεται, ε, μάλλον επιθυμείται, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές από μόνες του να αποφασίσουν είτε την προστασία του περιβάλλοντος είτε τις τοπικές ανάγκες ανάπτυξης. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο που ελοχεύει, γιατί αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει αντίθεση μεταξύ των δύο και μια επιλογή που πρέπει να γίνει ει βάρο του περιβάλλοντο όμω. Και αυτό, σε αυτό ευχαριστώ την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Υπενθυμίζω ότι θα ψηφίσουμε, θα κατατεθούν τροπολογίες, αλλά αν χρειάζεται να συνεχιστεί η συζήτηση, ο κύριος Ματούλα είναι πρόθυμος να συνεχίσει και να τα ακούσει όλα τα σχόλια. Άλλα σχόλια υπάρχουν? Όχι. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Προτείνω να είναι η 3η Μαρτίου το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι. 12 τρίτου, ε, συγγνώμη, 3 τρίτου, 12 το μεσημέρι. Ε, καθυστέρησε λίγο να έρθει από την Κομισιόν στο Κοινοβούλιο Dirk Κάνερ, οπότε για να μην χάνουμε χρόνο ας πιάσουμε κι άλλη γνωμοδότηση και αν χρειαστεί θα διακόψουμε. λοιπόν, να αρχίσουμε. Το σημείο 10 είναι ο κύριος Σάνερ. Το προσπερνάμε προς το παρόν, πάμε στο 11 που είναι η Ένωση Καινοτομίας μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για ένα κόσμο μετά την κρίση. Ε, δεν ενδιαφερόταν κανείς αν θυμάστε και ανέλαβα εγώ τη γνωμοδότηση. Για να προετοιμάσω την πρόταση και αυτό που θεώρησα ότι ήταν σημαντικό και έπρεπε να προσθεθεί στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ήτρε είναι ακριβώς αυτό για το οποίο είμαστε αρμόδιοι, δηλαδή την περιφερειακή διάσταση της πολιτικής καινοτομιών και την εφαρμογή της πολιτικής καινοτομιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Και ακριβώς εδώ πρέπει να τοποθετήσουμε την καινοτομία που είναι ένα σύνδεσμος μεταξύ ερευνητική κοινότητα και επιχειρηματικής κοινότητα, ε, όπου η ε, σύνδεση αυτή θα είναι πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Προτείνω λοιπόν να προσθέσουμε στη γνωμοδότηση της ΙΤΡΑ, της Επιτροπής Βιομηχανίας, ε, να προσθεθεί λοιπόν αυτό το περιφερειακό επίπεδο όπου η διαδικασία των καινοτομιών θα πρέπει να στοχεύει και να εστιάζει. Θα πρέπει Εκεί δηλαδή να αναφερθούμε στην υποδομή και την ικανότητα ε, φαρμογής μιας καινοτόμου προσέγγισης της ανάπτυξης. Θέλω επίσης η γνωμοδότησή μου να αναφέρεται και στην ευθύνη των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο να γνωρίζουν πολύ καλά ακριβώς ότι το περιφερειακό επίπεδο μπορεί να αναπτυχθεί και να αναπτύξει καινοτόμους δραστηριότητες και επίσης τονίζω το γεγονός ότι και οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινότητες που δεν έχουν πανεπιστήμια ή κέντρα έρευνας δεν θα πρέπει να δημιουργούν, να παράγουν γνώση για να είναι καινοτόμα, μπορούν να, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις περιφέρειες και τις ε, τοπικές κοινότητες που δεν έχουν πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα να αναπτύξουν και εκείνες το καινοτόμο δυναμικό τους. Επίσης αναφέρομαι στη σημασία των μη τεχνολογικών καινοτομιών γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα σε περιφερειακό ακριβώς και τοπικό επίπεδο όπου υπάρχουν ένα σωρό βέλτιστες πρακτικές σε αυτό το τομέα και επίσης αναφέρομαι στις συζητήσεις που κάναμε για τις περιφερειακές πολιτικές και τις καινοτομίες και σε αυτά τα πλαίσια ε, υπογραμμίζουμε, υπογραμμίζουμε την ανάγκη εντοπισμού κοιμόμενων καινοτόμων που ακούσαμε τόσες φορές να αναφέρονται στις ακροάσεις που οργανώσαμε και ενθαρρύνω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει περαιτέρω βήματα για την ε, δημιουργία χρηματοδοτικών μηχανισμών, ιδιαίτερα σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά ε, δημοσιονομικά όργανα υπεύθυνα για τον προϋπολογισμό, ούτω ώστε να βελτιωθεί η μόχλευση στον τομέα των κοινοτομιών. Αυτά ουσιαστικά ήθελα να σας πω. Deadborn, Michael Troider. Α, εδώ είναι. Δεν τους βλέπω. Οι σκιώδεις λοιπόν είναι εδώ. Θέλουν να μιλήσουν. Α, Ελίζαμπετ, ε, δεν σε είχα σημειώσει. Ποιος ε, παίρνει πρώτο το λόγο. Η κυρία Σρότερ. Εγώ ε, δεν ξέρω αν έχει δηλωθεί αυτό, αλλά είμαι σκιώδης. Είναι καλό, καλό το κείμενο και γνωρίζω και τη συζήτηση σε άλλες επιτροπές για αυτό το θέμα. Λείπει κάτι άλλο ε, που το ζητάμε σε άλλες περιπτώσεις, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση δηλαδή. Περιφερειακές καινοτομίες, δεν είναι σαφές εκεί όμως ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουν οι καινοτομίες, ενώ νομίζω ότι αυτό αποσαφηνίζεται στο έγγραφο της Κομισιόν. Και επίσης μου αρέσει η ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, που θα διασφαλίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Κάποιες ε, καινοτομίε δημιουργούν και θέσεις εργασίας και αυτό πρέπει να το τονίσουμε γιατί αυτό θα δώσει όθηση για να εφαρμοστούν αυτές οι καινοτομίε και με τη βοήθεια των διαρθρωτικών ταμείων, γιατί αυτό θέλουμε σε τελευταία ανάλυση. Να πούμε, αν χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία, θα πρέπει αυτό να έχει νόημα στα πλαίσια της ε, ε, ολοκληρωμένης προσέγγισης, να ωφελεί την περιφέρεια, να διασφαλίζει ε, αυξημένη απασχόληση και αηφορία βέβαια, διατηρησιμότητα. Αυτά λείπουν λίγο. Είναι λίγο υπερβολικά τεχνική η έκθεση αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει καινοτομία, Υπάρχουν προτάσεις για την καινοτομία, αυτά τα λέει, χωρίς όμως να επισέρχεται στα κεντρική σημασίας θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Γιατί αυτό θα είναι προτεραιότητα για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πώς θα διαμορφώνονται όλες αυτές οι δραστηριότητες, ούτως ώστε αν υπησέλθει το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τότε όντως να εξυπηρετούνται οι στόχοι της Ευρώπης 2020. Ε, και θα φροντίσω μέσα από τροπολογίες να το καλύψω αυτό. Πολύ σύντομα, η καινοτομία είναι ένα θέμα που είναι ε, πολύ σημαντικό στα διάφορα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια και, την Κομισιόν. Και περιμένουμε ε, στοιχεία από την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη ε, να προωθηθούν και από τον αρμόδιο επίτροπο. Και πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν γιατί η καινοτομία και η ε, ανάπτυξη έχουν ε, μεγάλη ε, διασπορά θα έπρεπε να εστιαστούν περισσότερο και στο περιφερειακό επίπεδο και οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές έχουν τεράστιο ρόλο να παίξουν εδώ. Νομίζω το ερώτημα είναι πώς θα ενθαρρύνουμε αυτές τις διαδικασίες δημιουργώντας μηχανισμούς ώστε να λάβουν χώρα. Έχουμε και εμείς το ρόλο μας να παίξουμε, αλλά θα πρέπει να γίνει συζήτηση και με τα θεσμικά όργανα, για παράδειγμα την Επιτροπή των Περιφερειών, που είναι πολύ σημαντικός παράγων ε, Ενεργοποίηση των περιφερειών για τέτοιε δραστηριότητε στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Σαγκουράκης. Ναι, δύο μικρά σχόλια κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να σα παρακαλέσω να διευκρινίσετε όταν αναφέρεστε σε μη τεχνολογικέ έρευνες τι ακριβώ εννοείται. Και εγώ συμφωνώ, αλλά πάντω να δούμε τι, τι ακριβώς είναι αυτό οι μη τεχνολογικέ έρευνες. Και ένα δεύτερο, έχω ξέρετε μια γενικότερη ένσταση ή μάλλον έχω την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε ένα γενικότερο ερώτημα. Νομίζω, όπως και εσείς, ότι η Επιτροπή μας είναι εδώ για να βοηθήσει τις περιφέρειες να αναπτυχθούν, να κατακτήσουν ένα πιο ψηλό επίπεδο ανάπτυξης από αυτό που έχουν τώρα. Και αυτό είναι και περιφερειακή ανάπτυξη η Επιτροπή μας. Έχω όμως τη γνώμη ότι η ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας στις περιφέρειες δεν οδηγεί κατά ανάγκη σε αυτό το στόχο. Δηλαδή μπορεί να έχετε μέσω μιας πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας δημιουργία center of excellence όπως λέγονται, πολύ υψηλού επίπεδου ερευνητικά κέντρα σε κάποιες περιοχές οι οποίες γενικά όμως δεν είναι πίσω από οικονομική ανάπτυξη. Έχω τέτοια παραδείγματα στην Ελλάδα, έχω και αλλού. Άρα το ζητούμενο για μας είναι πώς τα αποτελέσματα της έρευνας και της τεχνολογίας θα συνδεθούν με τις ανάγκες ανάπτυξης συγκεκριμένων περιφερειών και όχι γενικά η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας. Δεν οδηγεί γενικά δηλαδή η ανάπτυξη τη έρευνα και της τεχνολογία σε μια περιοχή στην ανάπτυξή τη. Και αυτό το ζήτημα το έχω θέσει και άλλη φορά στην Επιτροπή. Δεν υπάρχει απάντηση στο ζήτημα αυτό και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Για δύο λόγους. Γιατί καταρχήν δεν νομίζω ότι η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση στους στόχους της έρευνας και της τεχνολογίας βάζει αυτά που έχουν πραγματικά ανάγκη οι εργαζόμενοι, αλλά είναι οι ανάγκες κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων. Και δεύτερον, πολύ πιο σημαντικό, ακόμα και αυτή η έρευνα δεν συνδέεται με την παραγωγή. Δεν συνδέεται με την παραγωγή ούτε στην Πολωνία, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ιταλία. Αλλά αυτό που γίνεται τι είναι. Η έρευνα της Ελλάδας συνδέεται με την παραγωγή της Γαλλίας και η έρευνα της Πολωνίας με την παραγωγή της Αγγλίας και ανάποδα. Γι' αυτό το λόγο κιόλα, εάν δεν λυθεί το πρόβλημα που σας είπα κυρία Πρόεδρε, που δεν είναι κατά ανάγκη και θέμα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, αλλά είναι δεχομένω χρήση τεχνολογιών για την ανάπτυξη των περιφερειών, δεν θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Any other comment? Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα σχόλια, παρακαλώ. Εν συντομία για να απαντήσω στο ερώτημα σα. Νομίζω θα απαντήσετε εσεί ο ίδιο στο ερώτημά σα όταν ρωτήσατε στην αρχή τι σημαίνει non-technological innovation και είπατε δηλαδή ότι δεν μπορείτε να υποθέσετε ότι κάθε περιφέρεια, κάθε περιοχή θα πρέπει να αναπτύξει δηλαδή την έρευνά της και νέες τεχνολογίες να τις αξιοποιήσει. Αυτό που προσπαθώ να πω δηλαδή είναι το εξή. Μπορεί να είσαι ιδιαίτερα καινοτόμο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρέχει μια υπηρεσία, μια δημόσια υπηρεσία χωρίς να υπάρχει αν θέλετε κανένα input νέων τεχνολογιών. Μπορείς επίσης να ασκείς με καινοτόμο τρόπο την ε, διεύθυνση θέλετε, της επιχείρησής σου. Καινοτομία δεν σημαίνει αναγκαστικά και μόνο δηλαδή, αν θέλετε μια έρευνα δηλαδή η οποία και τεχνολογική βάση. Υπάρχουν ε, ιδιαίτερα επιτυχή παραδείγματα περιφερειών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Σε όλη την Ευρώπη. Στη Φιλανδία Φερρυπίν μπορείτε να βρείτε τις περισσότερες από αυτές, οι οποίες δεν έχουν, αν θέλετε, ούτε ερευνητικά κέντρα, αλλά ούτε και την απαραίτητη γνώση εκεί, αλλά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Κάνουν τα πράγματα διαφορετικά δηλαδή από ό,τι συνείδησαν να κάνουν, προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση, σε να προσελκύσουν νέους, να έρθουν και να μείνουν εκεί. Αυτό προσπαθώ να πω δηλαδή και εγώ, ότι πρέπει να την εννοήσουμε την ε, καινοτομία έτσι με τον ευρύτερο τρόπο. Όχι αντισυνδέατο με την έρευνα δηλαδή αναγκαστικά, αλλά αν είσαι καινοτόμο δηλαδή, απαντώντα αν θέλετε στα αιτήματα και ικανοποιώντα τι ανάγκε αν θέλετε των ανθρώπων με τρόπο διαφορετικό από ό,τι στο παρελθόν. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η ενθάρρυνση των περιφερειών για το πώ θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικέ και καλύτερε σε αυτό που κάνουν, χωρί δηλαδή να μπλεχτούν, να θέλετε, με νέε τεχνολογίε ή να αξιοποιήσουν, αυτά τα πρόσφατα αποτελέσματα τη έρευνα. Ε, πάντως σας κατάλαβα αυτό που είπατε, όσον αφορά τι μη τεχνολογικέ καινοτομίε, και βρισκόμαστε εδώ για να αποφασίσουμε για την προθεσμία Υποβολή τροπολογιών. Δυστυχώ ε, το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι πολύ σύντομο, άρα υπάρχει αυτό ο περιορισμό και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, αλλά η προθεσμία είναι 3 Μαρτίου δηλαδή, το μεσημέρι και πάλι, 12 το μεσημέρι. Σημείο 10 τώρα τη ημέρη τη διάταξη, σα πάμε πίσω δηλαδή, που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ντυρικάνερ, ο οποίο είναι Γενικό Διευθυντή Περιφερειακή Πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε να μα πείτε, κύριε Άνερ, το πώ η πολιτική αυτή συμβάλλει στην ε, στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Τώρα με την τρέχουσα δηλαδή έκδοση της πολιτικής όπως και τη μελλοντική της έκδοση. και πώς θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε πώς από την μικής απόψεως προσαρμόζοντας αν θέλετε την τρέχουσα περίοδο στην ε, πολιτική για την Ευρώπη του 2020 πόσο ευέλικτοι είμαστε σήμερα Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή κάτι σχετικά με την καινοτομία μέσω της ε, πολιτικής αυτής για την Ευρώπη του 2020 ή κάποιες άλλες αυτές τις πρωτοβουλίες ναυαρχίδες. Αν είχατε περισσότερες πρακτικές πληροφορίες να μας δώσετε θα σας ευγνωμονούσαμε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλησπέρα σας και σας ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά σήμερα δημοσιεύθηκε μία έκθεση για το ανθρώπινο κεφάλαιο και την περιφερειακή διάσταση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ήμουν σε μία στρογγυλή τράπεζα για το θέμα αυτό, γι' αυτό και καθυστέρησε. Θα ήθελα να σας αναφέρω τα πολιτικά συμπεράσματα αυτή τη έκθεση που περιοριζόταν σε κάποιου δείκτε και πιο τεχνικά θέματα. Πάντω, τα πολιτικά συμπεράσματα τη έκθεση ήταν ότι οι περιφέρειες πολύ περισσότερο από ότι οι ίδιες οι χώρες είναι αυτές που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία μιας στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό. Και μάλιστα καθορίζουν ακόμη και το 71% των διαφορών σε διαφορά τη δημιουργία πλούτου μεταξύ τους. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο ανθρώπινο δυναμικό, όπως είναι η στρατηγική του 2020, θα πρέπει να επικεντρώνεται στις περιφέρειες από την πλευρά τους οι περιφέρειες ε, θα μπορούσαν να συμμετέχουν πιο επικοδομητικά και να προταχθούν ως ε, ο πρωταρχικός και ο σωστός εταίρος για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ε, Ανάπτυξης. Αυτά είναι τα πολιτικά συμπεράσματα αυτής της έκθεσης που ούτως ή άλλως έχει επιβεβαιωθεί και μια τελείως διαφορετική ανεξάρτητη μελέτη που έχει γίνει με το δίκτυο των 130 πόλεων στην Ευρώπη και η δεύτερη έκθεση έδειξε ότι σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, αυτό που ενδιαφέρει είναι η περιφερειακή διάσταση και η τοπική διάσταση σε ορισμένε περιπτώσει. Και αυτή είναι πρωταρχική σημασία. Και μάλιστα ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι δύο τα δύο τρίτα των προσόντων και των δεξιοτήτων που έχουν σήμερα οι ε, ε, άνθρωποι τα, τις αποκτούν τις δεξιότητες αυτές και τα προσόντα στην, ε, στην ενήλικη ζωή τους. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το περιφερειακό πλαίσιο και στο πλαίσιο αυτό η σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Και σίγουρα αυτό είναι ένα από τα σημεία που θα πρέπει να έχουμε κατά νου συζητώντας για το μέλλον αυτών των πολιτικών μας. Επανέρχομαι τώρα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020. Είναι αλήθεια ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο και το κοινωνικό κεφάλαιο έχουν εξέχοντα ρόλο στην στρατηγική του 2020. Και οι αναπτυξιακές στρατηγικές για το ανθρώπινο κεφάλαιο θα αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά υπάρχουν και άλλα σημαντικά σημεία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020 και συνδέονται και αυτά με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι το θέμα της καλύτερης κοινωνικής ένταξης, το θέμα της καινοτομίας. Όλα αυτά εμπίπτουν στο κεφάλαιο της εφιούς ανάπτυξης, smart growth. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρούσα περίοδο, ε, μία παρατήρηση που κάναμε ε, με βάση τα έτη 2009 και 2010 είναι εξή. Καταρχήν θα θυμάστε ότι αυτή η διετία 2009-2010 ήταν η διετία της ε, σοβαρής κρίσης και το 2008 αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε σημαντικά με ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο ανατολισμό των πολιτικών μας και θα πρέπει και η πολιτική συνοχή να συμβάλλει στην ανάκαμψη. Αυτή η συνεισφορά χαρακτηρίστηκε από δύο βήματα. Η πρώτη Τη συμβολή ήταν το 2009 που επιτρέψαμε μια παράταση της εφαρμογής ε, της περιοδου 2000-2006 ε, κατά ένα εξάμεινο ώστε να προλάβουν τα κράτη-μέλη να εκταμιεύσουν ε, όσο περισσότερα κονδύλια είχαν απομείνει από την προηγούμενη περίοδο. Επίσης προστατεύσαμε να βελτιώσουμε τη ρευστότητα των κρατών μελών και για τη νέα περίοδο και προσπαθήσαμε επί τόπου να περάσουμε στην εφαρμογή της νέας περίοδου. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι μετά τον Ιούνιο του 2009 η εφαρμογή των πολιτικών επιτόπου εκτινάσεται στα ύψη. Και αυτό συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2010 σε πολλές χώρες μέλη και οδήγησε σε μια κατάσταση όπου είχαμε βέλτιστη χρήση του προϋπολογισμού του 2010 και χρήση για τις ε, ενδιάμεσες πληρωμές, δηλαδή για την αποπληρωμή δράσεων ε, που είχαν ήδη λάβει χώρα και προγραμμάτων που είχαν ήδη εκτελεστεί. Και όταν ε, βλέπουμε εκ του σύνεγγες αυτές τις δράσεις, διαπιστώνουμε ότι πολύ συχνά συνδυάστηκαν με μία μεταβίβαση των προγραμμάτων, όχι με επίσημες τροποποιήσεις των προγραμμάτων, αλλά ήδη εντός των προγραμμάτων υπήρχε περιθώριο λιγμών για τις χώρες και τις περιφέρειες, χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης, για να γίνει μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα και πολλές χώρες εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη δυνατότητα. Από τις αρχές του 2010 διαπιστώνουμε όλο και περισσότερες αλλαγές προγραμμάτων. Και αυτές οι αλλαγές των προγραμμάτων περιλαμβάνουν κυρίως δράσεις που ευθυγραμμίζονται και με τη στρατηγική του 2020. Ένα παράδειγμα που αν δεν έχει δημοσιευθεί, ελπίζω ότι θα δημοσιευθεί σύντομα, αφορά το θέμα της, των μέτρων της ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι μισές χώρες μέλη έχουν ήδη, οι περιφέρειες μάλλον των, των μισών χώρων μελών, έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας και από ό,τι ξέρω στη Γαλλία θα πρέπει να το ελέγξω όμως, σχεδόν ε, όλες οι περιφέρειες είναι, έχουν φτάσει στο όριο του 4%. Θα το ελέγξουμε πάντως. Αυτό που φαίνεται είναι ότι οι περιφέρειες αρχίζουν και λαμβάνουν υπόψη της και εφαρμόζουν και εμπράκτος τις νέες δυνατότητες των πολιτικών. Και πολλές περιφέρειες, και μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, είχαν από πριν προγράμματα που ευθυγραμμίζονταν σχεδόν απόλυτα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερος γιατί και αυτά τα προγράμματα προχωρούν και προοδεύουν. Λίγες περιπτώσεις έχουμε με προγράμματα που έχουν καθυστερήσει και εκεί θα πρέπει τους επόμενους μήνες να επενδύσουμε περισσότερο ώστε να σημειωθεί πρόοδος και σε αυτά. Γενικώ πάντως ήθελα να πω ότι φαίνεται καταρχήν ότι κατορθώσαμε να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας ό,τι αφορά τη συμβολή μας στην ανάκαμψη και την έξοδο, διέξοδο από την κρίση, χάρη στις επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχή, αυτό είναι το ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, παρατηρούμε σε πολλές χώρες μέλη και περιφέρειες κάποιες αλλαγές ή μεταβολές προγραμμάτων προκειμένου αυτά να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με την στρατηγική του 2020. Επίσης, σίγουρα θα συμφωνούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν μείνει πίσω, κάποιες περιφέρειες που υστερούν και θα πρέπει να αντισταθούμε αυτή την τάση ε, και να μείνει καινοτομία στην θεωρία. Θα πρέπει να την μεταφέρουμε και στην πράξη. Πάντως η γενική εντύπωση από τη διετία 2009-2010 είναι πολύ θετική κατά τη γνώμη μου. Τώρα, ερχόμαστε στην περίοδο μετά το 2013 για την περίοδο αυτή δύο, τα, δύο πράγματα είναι τα πιο σημαντικά. Πρώτον, τι μπορούμε να κάνουμε ήδη από τώρα για να προετοιμάσουμε κάποιους, κάποιους διάβλους για τις νέες γενναίες προγραμμάτων. Να προλιάνουμε το έδαφος και για τα νέα προγράμματα. Ήδη από το φθινόπωρο και με τις περιφέρειες που είναι πρόθυμες και με τις ε, χώρες μέλη που ενδιαφέρονται θα αρχίσουμε συζητήσεις για το πώς θα δημιουργήσουμε αυτά τα project pipelines και πώς οι εθνικές και περιφερειακές ε, στρατηγικές μπορούν να αναπτυχθούν ώστε να αξιοποιήσουμε το χρόνο και να μην χάσουμε καθόλου χρόνο να γίνεται ε, από τη μετάβαση στη, από την παλιά στη νέα περίοδο του 2014. Ήδη έχουμε διάφορους μηχανισμούς διαβούλευσης όπως το μηχανισμό Jaspers και τώρα θα πρέπει να δούμε αν τα περισσότερα προγράμματα αυτής της περίοδου έχουν περάσει από το Jaspers. Γιατί θέλουμε αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει το Jaspers να τη χρησιμοποιήσουμε για να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες ε, να έχουν διαβούλευση μέσω του Jaspers για την προετοιμασία και κατάρτιση προγραμμάτων για τη νέα περίοδο. Και να δούμε κατά πόσο υπάρχει ανάγκη εκ μέρους κάποιων χωρών για βοήθεια σε ό,τι αφορά τη δημιουργία των project pipelines. Αλλά αυτό θα το δούμε επί τούτου. Δεύτερο σημείο είναι το νομικό πλαίσιο. Και πώς θα έχουμε και μια νομική πτυχή της στρατηγικής του 2020. Πώς θα μεταφέρουμε τη στρατηγική του 2020 και σε ένα νομικό πλαίσιο. Οι αρχές εδώ είναι απλούστατες. Η πρώτη αρχή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020 ως πολιτικό όραμα η όραμα πολιτικών είναι υπερβολικά γενική και αόριστη και δεν επιτρέπει τη δημιουργία κάποιων επενδυτικών προτεραιοτήτων για την στρατηγική του 2020. Γι' αυτό και προσπαθούμε αυτή το, αυτόν τον ευρύ στόχο του 2020, της στρατηγικής του 2020, να το μεταφέρουμε στρέψουμε σε πιο συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες και σε συγκεκριμένους τομείς. Προσπαθούμε να εστιαστούμε σε τομείς και να προσελκύσουμε ε, τις ε, χώρες και τις περιφέρειες σε αυτούς τους τομείς προκειμένου να επιλέξουν τις προτεραιότητές τους για την επόμενη περίοδο. Και θέλουμε οι περιφέρειες και οι χώρες μέλη να σταθούν σε, σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει κάποια ελαστικότητα στο σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας, αλλά καλό θα ήταν να περιοριζόμαστε σε συγκεκριμένε σε λίγες προτεραιότητες. Αυτό θα προσπαθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ελπίζω ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 2011 θα είμαστε σε θέση να σας υποβάλουμε το νομικό πλαίσιο. Πάντως, ο στόχος μας, ο χρονικός μας ορίζοντας αυτή τη στιγμή είναι να το έχουμε έτοιμο για το φθινόπωρο αυτό το νομικό πλαίσιο. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι στην επόμενη περίοδο με αυτό το ευρύ νομικό πλαίσιο ως υπόβαθρο θα εξετάσουμε την κατάσταση σε κάθε χώρα μέλος και στις περιφέρειες της κάθε χώρας για να δούμε πώς ε, έχει κατάσταση σε κάθε χώρα και περιφέρεια και ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτεραιότητες ή οι τομείς προτεραιότητας ε, που θα τραβήξουν την προσοχή των περιφερειών. Μερικές φορές ε, μεταξύ των περιφερειών ίσως υπάρχουν διαφορές γιατί άλλες προτεραιότητες θα έχει για την επένδυση η Βόρεια Σουηδία από την Νότια Σουηδία. Ακόμη και στην ίδια χώρα δηλαδή οι περιφέρειες μπορεί να επικεντρωθούν σε διαφορετικές προτεραιότητες ή τομείς προτεραιότητες. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ελαστικότητα ώστε κάθε περιφέρεια να προσδιορίσει το κέντρο του ενδιαφέροντός της. Αλλά χρειαζόμαστε μια τέτοια εστίαση, γιατί όσο πιο ευρύ είναι το πρόγραμμα, τόσο περισσότερες προτεραιότητες μπορεί να καλύψει και θα πρέπει από κοινού τα κράτη-μέλη να προσδιορίσουμε όχι στο έπακρο, όχι μέχρι τελευταίες λεπτομέρειες, ποια είναι η καλύτερη κατάσταση, η καλύτερη ευκαιρία για κάθε χώρα. Επίσης θα πρέπει να συμφωνήσουμε πώς θα παρακολουθήσουμε από κοινού την πρόοδο και πώς θα καταμετρήσουμε την πρόοδο με βάση αυτούς τους τομείς προτεραιότητες και σε κάθε χώρα θα δούμε αν ε, υπάρχουν οι παράγοντες επιτυχίες για να επιτρέψουν την ευόδοση του προγράμματος. Χρησιμοποιούμε συνήθως τον όρο αιρεσιμότητα ή όρη. Εγώ προτιμώ να μιλάω για παράγοντες επιτυχίας. Γιατί με βάση την εμπειρία μας από την τρέχουσα περίοδο διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, να ισχύουν όροι για να έχουν απόδοση οι επενδύσεις. Όταν έχουμε μία σημαντική επένδυση στον περιβαλλοντικό τομέα, για παράδειγμα, στο νερό, για παράδειγμα, για την διαχείριση λιμάτων ή το πόσιμο είδωρ, από τη στιγμή που θα προβλεφθούν οι επενδύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από τον πληθυσμό. Θα πρέπει να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο να υπάρχουν οι διατάξεις αλλά και το σωστό σύστημα αποτίμησης ή υπολογισμού του κόστους. Επίσης, όταν έχουμε την καινοτομία ως προτεραιότητα επενδυτική και πάλι χρειαζόμαστε μία συνεκτική στρατηγική καινοτομία για τη χώρα και τις περιφέρειές της. Ορισμένα από αυτά τα θέματα είναι ζητήματα κοινή συλλογική, αλλά και πάλι δεν ε, συντρέχουν πολλές φορές. Γι' αυτό αναλύουμε την κατάσταση ανά όρο, ανά παράγοντα, σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια, ώστε όταν διαπιστώσουμε ότι κάπου υπάρχει ένα έλλειμμα που δεν συντρέχει μια προϋπόθεση, να μην είναι αυτό αποτρεπτικό για να μην επενδύσουμε, αλλά τη στιγμή που κάνουμε τη διάγνωση του ελλείμματος, να φροντίσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Ένα άλλο κεφάλαιο που βλέπω στη συμφωνία με τα κράτη-μέλη αφορά το συντονισμό, αυτό το κεφάλαιο, όπου πρέπει να φροντίσουμε καλύτερα από ότι σε αυτή την περίοδο, για να τα λέμε και σωστά, πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν καλύτερα να λειτουργούν δύο είδη συντονισμού. Πρώτον, συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ε, μέσων κοινοτικών, ενωσιακών. Δεύτερον, μεταξύ συντονισμός μεταξύ ενωσιακών και εθνικών μέσων και συστημάτων επενδύσεων. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί από την αρχή και θα είναι κομμάτι αυτού που λέμε Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, Σύμπραξης και ε, το συμβόλαιο συμπράξεων. Θεωρώ ότι θα πρέπει σε αυτά τα πλαίσια να υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις πρώτον εις ό,τι αφορά το συμβουλευτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, βοηθήσει αυτές τις καλές στρατηγικές ή τι μπορεί να κάνει για να φέρει σε επαφή η Κομισιόν κάποιες περιφέρειες με κάποιες άλλες, ώστε να μάθουν μεταξύ τους και να ωφεληθούν. Πολλά πράγματα μπορούμε να ε, θεωρήσουμε δεσμεύσεις που θα αναλάβει η Κομισιόν στα πλαίσια μιας τέτοιας συμφωνίας με ένα δεδομένο κράτος μέλος, για να γίνουν κάποια πράγματα. Και το μεγάλο πλεονέκτημα που βλέπω εγώ στην προσέγγιση αυτή, σε σύγκριση με μια προσέγγιση ή σε αντιπαράθεση με μια προσέγγιση όπου προσπαθούμε όλα να τα βάλουμε μέσα σε ένα γενικό κανονισμό, είναι ότι θα είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι και πολύ πιο εξειδικευμένοι σε επίπεδο εθνικό ή και περιφερειακό. Θα λαμβάνουμε τις ιδιαιτερότητές τους καλύτερα και θα γινόμαστε πιο κατανοητοί από τους πολίτες αυτής της χώρας, αφού θα αντιμετωπίζουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα τα δικά τους και όχι κάποια αφηρημένα προβλήματα που υποτίθεται ότι θα λύσουν ένα πρόβλημα. Γιατί ένα πρόβλημα στην Κρήτη, ας πούμε, μπορεί να μην γίνει καθόλου κατανοητό στη Βόρεια Φιλανδία. Θα υπάρχει δυνατότητα λοιπόν, προφανώς μέσα σε κάποιο νομικό πλαίσιο το οποίο θα είναι δεδομένο και θα υπάρχει, θα υπάρχει η δυνατότητα στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών εταιρική σχέσης να είμαστε πιο συγκεκριμένοι να εξειδικεύουμε τα σημαντικά και το επόμενο βήμα αφού θα υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες εταιρική σχέσης ε, μετά θα καταρτιστούν επιχειρησιακά προγράμματα. Εδώ δεν βλέπουμε μεγάλες αλλαγές σε σχέση με αυτά που γίνονται στην τρέχουσα περίοδο. Αλλά πρέπει να πω ότι μετά από πολλές συζητήσεις που κάναμε με τις περιφέρειες, με τα κράτη-μέλη, με συναδέλφους από τα κράτη-μέλη και με εσά επίσης, αναρωτιέμαι, και αυτό είναι προσωπικό δικό μου θέμα, αναρωτιέμαι πάντως, δουλεύω με 100% σωστά αφού παρατηθήκαμε από τα πολυταμιακά προγράμματα αυτή την περίοδο και έχουμε μόνο, μόνο ταμιακά προγράμματα. Γιατί αυτό στην πράξη μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα. Γιατί όταν είμαστε σε μια περιφέρεια και θέλουμε ανάπτυξη, έχουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο ας πούμε φέρνει, συνενώνει όλες τις ε, πηγές μαζί. Ε, αυτό είναι ας ένα έναυσμα για προβληματισμό, τροφή για σκέψη. Γιατί και εσείς μπορεί να βοηθήσετε και εμένα και τους συναδέλφους μου να τα σκεφτούμε καλύτερα τα πράγματα. Και έτσι περνώ στο τελευταίο θέμα μου. Πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά σε αυτή την τελική φάση. Καταρχήν θα αξιοποιήσουμε τις επόμενες εβδομάδες για να κάνουμε πάλι μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων με τους σημαντικότερους εταίρους για να βεβαιωθούμε ότι δεν παραβλέψαμε κάτι το σημαντικό εις ό,τι αφορά την απλοποίηση. Θα συναντηθούμε πάλι, θα οργανώσουμε συνάντηση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους τους εδώ. Θα οργανώσουμε συναντήσεις με συναδέλφους από τα κράτη-μέλη που εργάζονται στον τομέα αυτό, συναδέλφους από τις περιφέρειες που δουλεύουν επί τόπου, από τις ε, διαχειριστικές, τις ε, ε, αρμόδιες αρχές. Οπότε να μην παραβλέψουμε τίποτα και όλα να τα λάβουμε υπόψη μας εξακολουθούμε να συνεργαζόμεθα με την ομάδα υψηλού επίπεδου και έχουμε και μια ειδική ομάδα task force για την αιρεσιμότητα ή για τις προϋποθέσεις ε, ε, όπου εκπροσωπείστε και θα συζητήσουμε και με τους συναδέλφους από τα κράτη-μέλη και, την Επιτροπή των και στην Επιτροπή των Περιφερειών προσπαθούμε να διευκρινίσουμε αυτή την έννοια της αιρεσιμότητας ή της διατύπωσης προϋποθέσεων και τι ρόλο θα παίζει στην εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. Αυτά δουλεύουν τώρα επί τόπου. Εγώ ε, περιμένω τον Ιούνιο και αυτό δεν είναι καινούριο για σας την πρόταση της Κομισιόν για το δημοσιονομικό πλαίσιο και σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό θα πρέπει να εγκριθεί από την Κομισιόν με τον κανονισμό μας ε, τον Ιούλιο. Ελπίζω ότι θα γίνουν πράξη όλα αυτά και ελπίζω ότι θα δουλέψει το χρονοδιάγραμμα. Εμείς τουλάχιστον δουλεύουμε με τρόπο τέτοιο ώστε να τα προλάβουμε και τον Ιούλιο να τεθεί επιτάπητος και τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, όπως είπα, θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σε εθελοντική βάση με τις χώρες ή τις περιφέρειες, γιατί ακόμη δεν έχει λάβει απόφαση το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα. Θα αρχίσουμε λοιπόν συζητήσεις με τις περιφέρειες για να δούμε πώς βλέπουν εκείνες την επόμενη προγραμματική περίοδο πολύ συγκεκριμένα και επιτόπου σε σχέση με την Ευρώπη 2020. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι σε πρώιμη φάση και έγκαιρη φάση θα γίνει προετοιμασία των έργων, ώστε όταν εγκριθούν οι κανονισμοί να χρειαστεί ο πραγματικά ελάχιστος απαραίτητος χρόνος για τις τυπικές διαδικασίες. Αυτή είναι η προοπτική, το χρονοδιάγραμμα και τώρα περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις δικές σας αντιδράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ντύρκ. Βεβαίως και θα ακούσεις και από εμά αντιδράσει. Ο Λάμπερτ Βανίστελ Ρο είναι ο πρώτο. Ευχαριστώ που ήρθατε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Χαιρόμαστε που ήρθατε. Ε, κάναμε μια συζήτηση για την ε, έκθεση του Αντιπροέδρου κυρίου Σταυρακάκη, Αντιπροέδρου της Επιτροπής και κρίμα που δεν είναι εδώ γιατί νωρίτερα συζητήσαμε για τη μονοταμιακή προσέγγιση στη χρηματοδότηση των έργων και εσείς τώρα σε αυτό αναφερθήκατε. Πρέπει να ξανασκεφτούμε το μοντέλο. Αν δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ε, για τα ταμεία, το αλληλεία, το γεωργίας, ε, κοινωνικό κλπ. θα πρέπει να δίνει κάποιο όφελος, γιατί αλλιώς ε, δεν έχει κανένα νόημα. Αν είναι απόδοση. Είναι σαν να τραγουδούν παράφωνα πολύ μαζί. Τώρα λοιπόν η εδαφική διάσταση είναι σημαντική στη συνθήκη. Και εκεί γίνονται σύντονες προσπάθειες. Εμείς έχουμε ε, περιφερειακή προσέγγιση για το Περιφερειακής Ανάπτυξης Ταμείο και εθνική προσέγγιση για το Κοινωνικό Ταμείο. Δηλαδή άλλη γραφειοκρατία ασχολείται με το ένα και άλλη με το άλλο. Άλλη προσέγγιση για το ένα, άλλη για το άλλο. Αυτό είναι απορριπταίο. Άρα χρειάζονται μεγάλες αλλαγές. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να ξέρουμε ε, πώς, τι θα συζητήσετε με τα κράτη-μέλη. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, είδαμε ότι είναι πολύ συγκεντρωτική η προσέγγιση της κυβέρνησης και αν κολλήσουμε εκεί θα νομίζουμε ότι θα πετύχουμε τους στόχους της ε, Ευρώπης, ε, της στρατηγικής 2020, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα τα έχουμε κάνει καλά. Γιατί αν δείτε και το κοινοβουλευτικό ψήφισμα πριν από δύο εβδομάδες και τους στόχους 2020, θα δείτε ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ακόμα η διακυβέρνηση είναι αδύναμη. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα πολυεπίπεδα μέσα μας, αλλά με αποκεντρωμένη προσέγγιση θα χάσουμε σημαντικές ευκαιρίες. Η ερώτηση λοιπόν είναι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση όπως είπατε και εσείς με την πολυταμιακή προσέγγιση και έχουμε πιο έντονη ε, διαπεριφερειακή αν θέλετε ε, ε, συγκρότηση. Μπορεί να υπάρχουν και εδαφικές, εδαφικά σύμφωνα. Το 2011 θα Δεν γίνεται ε, από την αρχή να διατυπώνουμε τις ε, ε, λεπτομέρειες των εδαφικών οντοτήτων. Αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο θα αποτύχει. Μου έκανε εντύπωση αυτό που καταφέρατε τους τελευταίες τους τελευταίους μήνες και το κείμενο και το φόρουμ για τη συνοχή και το κείμενο του Συμβουλίου ήταν απόλυτα θετικό. Μπορείτε λοιπόν να μου πείτε ίσως το 2011 είναι το έτος της, ε, του στοχασμού που αρχίζει μετά και ο κανονισμός. Μετά το 2012 δεν φαντάζομαι να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στα προγράμματα γιατί πολλές χώρες έχουν ε, δεσμεύσει τα κονδύλια σε επιχειρησιακά προγράμματα. Στις κάτω χώρες δεν υπάρχει πολύ περιθώριο ελιγμών πια. Οπότε δεν πρέπει να περιμένετε και πάρα πολλά. Γιατί ήδη έχουν ληφθεί πολλές αποφάσεις για τα προγράμματα και τα έργα. Επίσης, αν έχετε ένα τέτοιο σύστημα διαπραγματεύσεων για τις συμβάσεις, μπορεί κάποια χώρα να πει, μάλιστα, θα λάβουμε υπόψη μας, ας πούμε, προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και άλλες μπορεί να μην το κάνουν. Ακόμα και για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Οι εμβληματικές δεν έχουν ακόμα τρέξει καλά. Η μία είναι για την ενεργό γύρανση ή την υγιή, ας γύρανση πώς θα γίνουν οι προσαρμογές αυτές τα επόμενα χρόνια. Μήπως παραείστε αισιόδοξο. Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρχει τόσο γρήγορη ανταπόκριση και σωστή και όλοι να καταλάβουν ας πούμε, τι κάνετε στα πλαίσια των εμβληματικών λεγόμενων πρωτοβουλειών. Ε, θα μας ενημερώσετε, 2011 αρχίζει ο κανονισμός, 2012 η πρώτη ανάγνωση και για να ε, συνεχίσει να παίζει το νομικό του ρόλο το Κοινοβούλιο, μπορεί στο ενδιάμεσο να εφαρμόζονται πολλά πράγματα καινούργια, γιατί μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην, στην χρηματοδότηση και σε πολλά άλλα. Δηλαδή, πώς θα τα μεθοδεύσετε όλα αυτά και πώς θα λειτουργήσουν στα πλαίσια του υφισταμένου κανονισμού. Ευχαριστώ που ήρθατε και ακούσατε τις ερωτήσεις μας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θαυμάζω την αισιοδοξία σας, κύριε Διευθυντά, παρόλο που δεν τον συμμερίζομαι. Δεδομένες της παρούσης καταστάσεως, τόσο στις χώρες της ζώνης ευρώ, όπως και στις υπόλοιπες, διότι μεταξύ του 2007 και του 2013, όπως όλοι μας γνωρίζουμε εξάλλου, στα κράτη-μέλη 270 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί και θα δοθούν. Και μας μένουν 134 δις ευρώ, τα οποία ακόμη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Η απορρόφηση δηλαδή μειώθηκε προοδευτικά και σταδιακά σε σχέση με την, περίοδο, την προηγούμενη περίοδο του προγραμματισμού. Αν στο παρελθόν δηλαδή, αν στο παρελθόν μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα κονδύλια αυτά χωρίς να είμαστε προσεκτικοί αν στο μακροοικονομικό σκέλος και στη μακροοικονομική πτυχή αυτών Σήμερα όταν πολλά κράτη-μέλη συνεχίζουν και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, μίσονες μάλιστα δυσκολίες, δεν επιτρέπουμε πλέον στον εαυτό μας την πολυτέλεια, δεν μπορούμε να μην ασχολούμεθα με την μακροοικονομική διάσταση. Του βεβαίω όσον αφορά τον πολιτικό και δηλωτικό χαρακτήρα, η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και οι στόχοι της είναι πάρα πολύ σημαντική ότι η πολιτική συνοχή παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην όλη αυτή υπόθεση. Όλοι συμφωνούμε προ αυτό και με αυτό. Πέραν όμω αυτού του δηλωτικού, αν και του πολιτικού χαρακτήρα, που πρέπει βεβαίω να λάβουμε υπόψη μα, διαφορετικά θα αργήσουν να φτάσουν τα αποθητά και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και εμείς το έχουμε πει, χωρίς, να ε, θεσπιστεί και να εφαρμοστεί αυτή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και ότι δηλαδή χωρίς να φτιάξουμε θέλετε αυτές τις ισότιμες σχέσεις εταιρικέ σχέσεις δηλαδή μεταξύ όλων δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πετύχουμε με την Ευρώπη και την στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Πρέπει κάτι να γίνει. Εγώ αρέσκομαι θέλετε στα συγκεκριμένα μέτρα, στα πρακτικά μέτρα. Και έχω κάποιε ερωτήσει, τα οποία ερωτήματα θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορούσε να μα απαντήσει και αν μπορεί να μα απαντήσει. Να ρωτήσω δηλαδή πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επεξεργαστεί έναν οδηγό ο οποίο θα απευθύνεται και θα έχει αν θέλετε ως παραλήπτες τις τοπικές και τι περιφερειακέ αρχέ που θα εξηγεί μέσα στον οδηγό αυτή την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την πρακτική αν θέλετε υλοποίηση και εφαρμογή αυτή τη αρχή, τη πολυεπίπεδη υλοποίηση. Γιατί χωρί αυτό, χωρί αυτόν τον οδηγό, μπορούμε να συμφωνούμε επί των αρχών και προ τι αρχέ, αλλά στην πράξη δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα. Τώρα, για το πρόγραμμα Έρασμος για τι τοπικέ και περιφερειακές αρχές, να πω κάτι. Συμφωνούμε όλοι, αλλά τίποτε δεν γίνεται. Τίποτε δεν συμβαίνει. Πράγμα αξιολείπητο. Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου έχουμε θέσει το ερώτημα αυτό με τις τροπολογίες που μου καταθέσει ή με τις ερωτήσεις που απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντα την ίδια θετική απάντηση λαμβάναμε και λαμβάνουμε, πράγμα το οποίο μα χαροποιεί μεν, αλλά δυστυχώς η αναμενόμενη απάντηση δεν την έχουμε ακόμη λάβει. Τι κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρακτικό επίπεδο. Σε λοιπόν το πρόγραμμα Έρασμου για τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ, ένα πρόγραμμα μεγάλη χρησιμότητα και το οποίο θα στηρίξει πραγματικά και θα μας βοηθήσει πραγματικά. Και ειδικότερα μια χρονική στιγμή όπου χρειάζονται αυτή την τεχνική βοήθεια οι τοπικέ και περιφερειακές αρχέ προκειμένου να βελτιώσουν, αν θέλετε, και την διοικητική του διαχειριστική του δυνατότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε ποτέ, αν μακρηγορείτε έτσι. Γιατί έχουμε δύο ακόμη εκθέσει για σήμερα και θα πρέπει να ορίσουμε την προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Και έχουμε και άλλου ομιλητέ. Αν όλοι μιλάτε λοιπόν για πέντε λεπτά, δεν θα έχουμε το χρόνο ούτε να ακούσουμε και τις απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Να θέσετε απλώς τι ερωτήσεις της. Παρακαλώ, κυρία Αντελή. Πρόεδρε, κύριε Χάινε, μιλήσατε αν θέλετε για το ανθρώπινο κεφάλαιο και αυτό έχει κεντρική σημασία το ανθρώπινο κεφάλαιο στην περιφερειακή του διάσταση είναι το πώς θα φροντίσουμε έτσι ώστε αύριο η ευημερία και η ποιότητα ζωής των πολιτών να βρίσκεται στο επίκεντρο των περιφερειακών πολιτικών. Καλό κάνατε λοιπόν και το υπενθυμίσατε. Υπενθυμίσατε επίση και είπατε ότι όντω υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία λειτουργούν καλά. Και το Urbac φέρει μια βέλτιστη πρακτική τα σχέδια αυτά, τα project αυτά, τα έργα αυτά θα πρέπει να ξαναβρούμε στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού γιατί λειτουργεί καλά και θα πρέπει να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Μιλήσατε κατόπιν για την ανάπτυξη. Προέρχομαι από την περιοχή Ile de France της Γαλλίας που είναι πολύ πλούσια αλλά πρόκειται για μια περιοχή όπου υπάρχουν αν θέλετε χειρότερες κοινωνικές ανισότητες. Θα πρέπει συνεπώς να ξαναδούμε το πώς βλέπουμε αυτή την ανάπτυξη και υπάρχει εδώ μια θέτηση σχέση αν θέλετε και για το ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά και τους δείκτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και να σχολιάσω κάτι έτσι εντάχει γιατί θα πρέπει να αφήσουμε τον χρόνο για τις απαντήσεις σας. Τη μεγάλη προτεραιότητα για τις ε, περιφερειακές πολιτικές πιστεύω που είναι αν θέλετε η ενεργητική αποδοτικότητα. Δύο μείζονες προκλήσεις κοινωνική πρόκληση και περιβαλλοντική πρόκληση πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και πρέπει συνεπώ να είμαστε θαραλέοι, τολμηροί γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε να επενδύσουμε και θα στοιχήσει πολύ ακριβά. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε το ζήτημα αυτό μακροπρόθεσμα για να σκεφτούμε δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα βεβαίω, αλλά και τις μελλοντικέ γενιές δηλαδή τα παιδιά σας και τα εγγόνια μας πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί ευθύ αμέσω να δούμε αν θέλετε τι γίνεται με την τεχνική βοήθεια γι' αυτό λοιπόν ήδη από τώρα Ας αναζητήσουμε, αν θέλετε, νέα αν θέλετε, χρηματοοικονομικά. Μην περιμένουμε το 2013, θα είναι πολύ πολύ αργά. Η επόμενη περίοδος προγραμματισμού, αν θέλετε, από τώρα πρέπει να ξεκινήσει. Τέλος, είπατε, ότι οι προϋποθέσεις θα θέλετε πραγματικής επιτυχίας στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που είναι, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αν θέλετε, όλοι οι παράγοντες. Μιλήσαμε προηγουμένως και μιλήσατε μάλλον προηγουμένως για την πολυεπίπεδη διάσταση αλλά ξανασκεφτείτε το ζήτημα τοπικά για να το δείτε και το ζήτημα αυτό αν θέλετε παγκόσμια. Να δούμε δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος των πόλεων σήμερα. Πώς είναι δυνατόν που υπάρχουν περιοχές στη Γαλλία που, που ορισμένες από αυτές φερρυπίν λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα περιερικά ταμεία ενώ άλλες όχι. Ένας από τους κινητήρες είναι να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό μακροπρόθεσμα αλλά με μια τοπική αν θέλετε διάσταση την οποία σήμερα δεν βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ξέρω την άποψή σα. Είπατε αφενό ότι κάθε κράτο θα πρέπει να έχει τι δικέ προτεραιότητε. Ναι, αλλά ποιο θα καθορίσει τα κριτήρια, εμεί ή τα κράτη-μέλη. Και ποια είναι τα κριτήρια. Κλιματικέ αλλαγέ, ε, οι κοινωνικέ ανισότητε, η πτώχεια κτλ. Όλα αυτά είναι σημαντικό και πρέπει να λέγεται. Συνεπώ τα κριτήρια θα πρέπει να είναι τα ίδια για του πάντε. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, να δούμε αν θέλετε ποια είναι οι, οι παράγοντες θα θέλετε, οι οποίοι θα πρέπει να τεθούν από κοινού προκειμένου να βρεθούν να θέλετε αξιόπιστες, διαρκείς, βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις. Και ευχαριστώ. Uh, thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ κύριε Στρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον ε, κύριο Γενικό Διευθυντή για την παρουσία του εδώ. Έχω όμως και μια ε, παρατήρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο της πέμπτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που αφορά στη στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ένα σημείο της έκθεσης, συγκεκριμένα στην παράγραφο 12, γίνεται λόγος για την ενίσχυση της στρατηγικής του προγραμματισμού μέσα από ενισχυμένη εταιρικότητα και στενό διάλογο μεταξύ κομισιών, κρατών μελών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, ανάλογα με την περίπτωση, as appropriate. Το κομμάτι αυτό που αναφέρει πως θα γίνεται αυτό όπου κρίνεται απαραίτητο, δηλαδή ανάλογα με την περίπτωση, αφήνει στην ουσία περιθώρια ώστε να μην είναι πλήρως δεσμευτικοί και υποχρεωτικοί οι κανόνες για την εταιρική σχέση. Εμείς θέλουμε να οριοθετηθούν ξεκάθαρα και με δεσμευτικά πλαίσια στα οποία θα μπορεί να αναπτυχθεί η εταιρική σχέση. Εσείς το θέλετε. Ευχαριστώ. Thank you, Marcus Piper. Ευχαριστώ, Μάρκος Πίπερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις και την προοπτική. Τώρα, για το conditionality, ε, τις μεταβλητές, ε, όπως το πούμε. Συμφωνώ γιατί αν δεν υπάρχουν λειτουργικές διαχειριστικές ε, παράμετροι θα κατασπαταληθούν τα χρήματα. Ε, και μετά θα δημιουργηθούν λύματα που θα ταλαιπωρήσουν τα κράτη-μέλη. Τώρα, για την ε, ε, επαλήθευση, εκθέσεις, επιβεβαίωσης, εδώ φοβούνται τα κράτη-μέλη μήπως δημιουργηθεί υπερβολική γραφειοκρατία. Δεν το έχω πολύ καταλάβει μέχρι τώρα το σύστημα. Από ό,τι κατάλαβα θα δώσετε, δίνετε υπερβολικές προϋποθέσεις στα κράτη-μέλη. Η διαπίστευση ας πούμε θα πρέπει να είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κάποιου ευρωπαϊκού φορέα, ο οποίος θα δίνει μια σφραγίδα και το, κράτη, το κράτος μέλος θα καταλάβει ότι αν διαθέτει αυτή τη σφραγίδα απαλλάσσεται από τη γραφειοκρατία. Θα έχει μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων. Αν παίρναγε αυτό το μήνυμα θα αυξάνεται και η αποδοχή του συστήματος. Αλλά το να... Ε, ή δεν κατάλαβα καλά. Δηλαδή αυτό που πάτε να κάνετε, να ελέγχουν τα κράτη-μέλη, αυτό δεν είναι σωστό. Τώρα, το, η στρατηγική 2020 και ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα. Είπατε ότι, ότι οι στόχοι της στρατηγικής 2020 είναι υπερβολικά γενικόλογα διατυπωμένοι και δεν μπορούν να λειτουργήσουν δείκτες συγκεκριμένοι. Τι θα κάνετε δηλαδή θα γίνει ας πούμε πάλι ένα earmarking, κάποια ε, δέσμευση ας πούμε ε, στο, στους στόχους 2020 ή θα υπάρχουν κάποιοι δείκτες που θα πείτε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και τους στόχους του 2020 και πάνω σε αυτή τη βάση θα δοθούν και τα κονδύλια. Τέλος, θα είναι ας πούμε σαν τη Λισαβόνα 85% δέσμευση κονδυλίων, earmarking, η πρικοδότηση αυτή ή θα υπάρχει ας πούμε μια δυνατότητα κρίσης και αξιολόγησης του προγράμματος για να συνεχίζεται η χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Κύριε Σαγκουράκης παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μια, μια διαπίστωση και μια ερώτηση στον κύριο Άνερ. Η πρώτη ε, διαπίστωση είναι ότι μέχρι στιγμής κανείς ούτε ο κύριος Σάνερ φυσικά, δεν μας έχει πείσει ότι η εκπλήρωση των στόχων Ευρώπη 2020 θα οδηγήσει σε σύγκληση της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν έχω διαβάσει καμία απόδειξη ότι αν υλοποιηθούν οι στόχοι του 2020, στο, μετά από 10 χρόνια οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι όλες στο ίδιο επίπεδο, για να μιλάμε για σύγκληση. Η ερώτηση όμως δεν έχει να κάνει με αυτό. Η ερώτηση έχει να κάνει με το εξή. Την έθεσε κάπως ο κύριος Βανίστεροι. Θα ξέρω κύριος Άνερ ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους διάφορα προγράμματα παλιότερα δεν έχουν υλοποιηθεί ή πρέπει να υλοποιηθούν. Όταν ο κύριος ε, Άνερ λέει ότι στο, μέσα στο 11 θα υπάρχει μια νομική βάση για τους στόχους 2020 και για την επιλεξιμότητα των προγραμμάτων και μάλιστα γίνεται λόγος για λίγα προγράμματα, για λίγους στόχους, ώστε να βλέπουμε το αποτέλεσμα. Όλοι θέλουμε αποτέλεσμα. Το ερώτημα μου είναι το εξή. Με τα παλιά προγράμματα τα οποία τρέχουν και οποία δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, τι θα συμβεί. Δεύτερη ερώτηση, εάν κατά την Κομισιόν στην επιλεξιμότητα θα είναι και προγράμματα και projects τα οποία δεν εμπίπτουν στη στρατηγική 2020 αλλά που αποδεδειγμένα μπορούν να συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη. Αυτά θα είναι επιλέξιμα ή θα μείνουν απ' έξω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. And the last question, Derek Vaughan. κύριος Derek Vaughan. Τελευταία ερώτηση. Πολλές συζητήσεις έγιναν στο παρελθόν για τη συμβολή στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020, και να επικεντρωθούμε σε ένα σημείο που ανέφερε και ο κ. Σάνερ, το σημαντικό θέμα της χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας ε, στη στέγαση. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα τμήματα του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης και θα ήθελα αυτό, αν γίνεται, να το επεκτείνουμε και στον επόμενο γύρο των διαρθρωτικών ταμείων και μετά το 2013. Στην Ουαλία, για παράδειγμα, περίπου 8.000 ε, νοικοκυριά επωφελήθηκαν από αυτό το πολύ επιτυχημένο σχέδιο. Να το επεκτείνουμε και πέρα του 2013 και ίσως να το επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς της στέγης. Για παράδειγμα, για να γίνουν κάποιες προσαρμογές ε, για το, για άτομα με ειδικές ανάγκες ή για ηλικιωμένους ανθρώπους ή για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ενοικιαστές γιατί πολλοί άνθρωποι που στηρίζονται στα κοινωνικά επιδόματα δεν μπορούν να βρουν ξανά το δρόμο στην αγορά εργασίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να επεκτείνουμε αυτό το μέτρο όχι μόνο πέραν του 2013 αλλά και σε άλλους ε, τομείς πέραν της στέγασης. Έχετε το λόγο κύριε Γενική Διευθυντά. Thank you very much, Mrs. Uh, Chair. Uh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τον κύριο Βανίστερο. Συμφωνώ ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να έχει και θετικό αντίκτυπο επί τόπου, στην πράξη και το τονίζω αυτό. Γιατί θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά εποφελούνται οι δικαιούχοι. Θα πρέπει να δούμε επιτόπου αν έχει αντίκτυπο το μέτρο που θεσπίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν περιφερειακά βλέπει κανείς το όφελος και χρειαζόμαστε μια εδαφική διάσταση. Και την εδαφική διάσταση θα πρέπει να τη δούμε συγκεκριμένα και θα εξαρτάται και από τα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και από το μέγεθος των περιφερειών ή των χωρών. Για ορισμένες περιφέρειες για ορισμένα προγράμματα, ίσως, ε, προβλήματα ίσως θα πρέπει να δούμε και το υποπεριφερειακό επίπεδο. Άλλες περιφέρειες ε, θα πρέπει να επιλύσουν τα προβλήματά τους μέσω ε, εθνικού επίπεδου και άλλες φορές έχουμε καλύτερη επίλυση των προβλημάτων σε διασυνοριακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο. Πάντως έχουμε και τους μηχανισμούς και τα προγράμματα που μας επιτρέπουν να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς. Στην επόμενη περίοδο καλό θα ήταν να δώσουμε έμφαση στην αποκεντρωμένη διαχείριση και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ε, και έρχομαι εδώ στο σχόλιο της κυρίας Μανέσκου ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι όταν επενδύουμε ότι το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που θέλουμε να αναμειχθεί όλο και περισσότερο στη διαδικασία ότι έχει αυτό το επίπεδο την απαραίτητη ικανότητα και το δυναμικό να διαδραματίσει όντω ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Βανίστερο, είπατε ότι παρά ήμουν αισιόδοξο για τις αλλαγές των προγραμμάτων. Είναι σαφές ότι σχεδόν όλα τα προγράμματα, με ελάχιστε εξαιρεσει ότι εφαρμόζονται. όλα σχεδόν τα προγράμματα εφαρμόζονται. Και μάλιστα μερικά προγράμματα ήδη έχουν κατανείμει το 90% των κονδυλίων τους. Για ορισμένα προγράμματα ακόμη δεν έχει γίνει πλήρης κατανομή. Και για ορισμένα προγράμματα έχει, έχουν κατανεμηθεί τα κονδύλια σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, αλλά διαπιστώνουμε εκ των υστέρων ότι η ζήτηση για τα προτινόμενα μέτρα στις προτεραιότητες αυτές είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Αυτό το διαπιστώνουμε και φέτος και κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε και το χρόνο. Θα πρέπει να γίνει μια επανεξέταση των αρχικών προγραμμάτων. Οπότε αναμένεται και περαιτέρω μεταβολή των προγραμμάτων. <clears throat> Αυτό που θα ήθελα να αποφύγουμε είναι αυτές οι αλλαγές των προγραμμάτων να μην πάρουν στραβό δρόμο. Δηλαδή, προσπαθώντας οπωσδήποτε να γίνει πλήρης εκταμίευση των κονδυλίων, να μην πέσει κανείς στην παγίδα και να αρκεστεί σε τομείς που δεν είναι τόσο σημαντικοί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων περιφερειών. Η σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ποιότητα και στους τομείς που καλύπτουν τα προγράμματα. Σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε πολύ δαπανηρές ε, επενδύσεις στις υποδομές και θα γίνουν αυτές όχι μόνο στην τρέχουσα περίοδο αλλά σίγουρα και στην επόμενη. Πάντως ε, ως γενικό κανόνα θα θέλαμε από κοινού με τις περιφέρειες να εξετάσουμε περισσότερο παράγοντες όπως επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, σε κοινωνικό κεφάλαιο, σε καινοτόμες προσεγγίσεις όχι κατά ανάγκη για να είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας και να έχουμε σε κάθε περιφέρεια και μια Silicon Valley, αλλά να αξιοποιούμε σε κάθε περίπτωση τις προηγμένες τεχνολογίες ή ε, μεθοδολογίες ή προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν αλλού ή που σχεδιάστηκαν και επινοήθηκαν αλλού να τις χρησιμοποιήσουμε και σε άλλο επίπεδο προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Και δεν έχω υπόψη μου κανένα πρόγραμμα στην περίοδο αυτή που να μην ε, χαρακτηρίστηκε από αυτή τη μέρημνα και από αυτή την επιθυμία να χρησιμοποιήσει την ανταγωνιστικότητα θα έλεγα και δεν είναι δόκιμος αυτός ο όρος εδώ, να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει το δυναμικό της κάθε περιφέρειας και να το βελτιώσει αυτό το δυναμικό στο έπακρο, προκειμένου να δώσει μια όθηση στην ανάπτυξη. Βέβαια, όθηση στην ανάπτυξη πολύ συχνά ε, γίνεται μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ε, διαφόρων περιφερειών. Κυρία Μανέσκου, αναφερθήκατε στο πρόγραμμα Έρασμος. Να σας πω ακριβώς που βρισκόμαστε με το Έρασμος. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πολύ καλό αυτό το πρόγραμμα και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούμε να εξακριβώσουμε είναι ποιο θα είναι το σημείο αφετηρίας μας. Να μην έχουμε ένα πρόγραμμα εράσμους ε, διακίνησης προς διάφορες κατευθύνσεις. Για δύο ε, λόγους, γιατί είχαμε ερετούς ε, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που πολλές φορές αντιμετωπίζουν περιορισμούς ε, στην πατρίδα τους και πρέπει κάποια στιγμή να βρίσκονται εκεί και ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε ήταν το θέμα της μετάφρασης και της διερμηνίας. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από έναν ε, τοπικό άρχοντα να ε, γνωρίζει κατά ανάγκη να μιλάει, να καταλαβαίνει ξένες γλώσσες, κοινοτικές γλώσσες. Και αυτό που θα κάνουμε ως σημείο φετηρίας λοιπόν, για να δώσουμε το εναρκτήριο λάκτισμα στη διαδικασία αυτή, είναι να έχουμε ένα είδος θερινού πανεπιστημίου χειμερινού πανεπιστημίου και τα δύο, οποία πανεπιστήμια θα προσκαλούμε πολίτες από διάφορες περιφέρειες και ε, δήμους και κοινότητες, ώστε να αφήνουν τη χώρα τους και να πηγαίνουν σε άλλο περιβάλλον, να συναντούν ε, συναδέλφους τους από άλλες χώρες και σε συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα, να λέμε σε μία εβδομάδα ας πούμε, όπου να έχουν τέτοιες ε, ανταλλαγές και επαφές με ομολόγους τους άλλων χωρών και εκεί να μαθαίνουν στοιχεία για την ε, χώρα που τους φιλοξενεί, που οργανώνει αυτό το πανεπιστήμιο, το χειμερινό ή το θερινό και τα δύο. Και νομίζω ότι έτσι θα δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου καταρχήν ένας ερετός θα μπορεί να συμμετέχει δύο και τρεις φορές σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και αυτές οι εκδηλώσεις ε, θα, τα θα τις χρησιμοποιήσουμε και για ανταλλαγή απόψεων και για καλύτερη ενημέρωση, για να μαθαίνει ένας από τον άλλον και για να φέρουμε σε επαφή τους ερετούς ε, μεταξύ τους και να μάθει ο καθένας πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διδάγματα και τις εμπειρίες των άλλων στο δικό του τοπικό επίπεδο. Από ό,τι ξέρω και με βάση το σχεδιασμό που έχουμε κάνει, αν πάνε όλα καλά, η διαδικασία αυτή θα αρχίσει το επόμενο έτος. Τον επόμενο χρόνο θα έχουμε το πρώτο θερινό πανεπιστήμιο στα τέλη Αυγούστου, γιατί το πλεονέκτημα είναι ότι η χώρα υποδοχής που οργανώνει αυτό το θερινό πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει και διαθέσιμα ε, δωμάτια, οι αιστείες, συνήθως στα πανεπιστήμια ισχύει κάτι υπάρχει δυνατότητα προσφοράς και καταλήμματος στον ίδιο χώρο που θα γίνονται τα σεμινάρια, οι συζητήσεις, οι τρογγυλές τράπεζες κτλ. Λοιπόν, τώρα θα είμαι λίγο σύντομος, αλλά έτσι κι θα τα ξαναπούμε τις επόμενες εβδομάδες. Η Ευρώπη 2020 αποτελεί πράγματι μια στρατηγική η οποία ρητά και εξάστερα περιλαμβάνει δηλαδή και τον, την κοινωνική συμπερίληψη. Στην ανάπτυξη αν θέλετε αυτή που περιλαμβάνει, που εγκλείει δηλαδή και υπάρχει μια σειρά μέτρων που πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο αυτό και εδώ και πάλι το ανθρώπινο κεφάλαιο και το κοινωνικό κεφάλαιο έχουν να παίξουν και παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και μια και πολύ συχνά τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να προσεγγιστούν παρά μόνο σε τοπικό επίπεδο ή σε μια μικρή περιφέρεια, Βεβαίω το τοπικό επίπεδο και οι πόλει ειδικότερα και κυρίω θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των κειμένων που γίνονται αυτή τη στιγμή θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, έχουμε την πρόθεση μάλλον να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τις πτυχές της τοπικής ανάπτυξης αλλά και της αστικής επίσης. Τώρα, για την εταιρική σχέση η προσέγγιση, κύριε Τρεμόπουλε, νομίζω ότι πρέπει να είναι δεσμευτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση και κάθε φορά θα χρειάζεστε πάντα τους ίδιους εταίρους για να δουλέψετε, αλλά νομίζω ότι όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης καταρχήν πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της συνολικής στρατηγικής και στον ορισμό της στρατηγικής. Και μετά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να δουλεύετε καλύτερα σε τοπικό επίπεδο, όπου θα πρέπει να προβλέπετε και η δυνατότητα να δουλέψει κανείς ε, με εταίρους στο τοπικό επίπεδο και άλλες φορές για να μπορεί να πρέπει να δουλέψετε σε μακροπεριφερειακό επίπεδο, για να πω ένα ακραίο παράδειγμα, με συνεργασίες. Πάντα όμως η προσέγγιση της εταιρικότητας μέσα από εταιρικέ σχέσεις είναι θεμελιώδης πυλώνας της πολιτικής μας ίσως να είναι και το μεγαλύτερο ε, πλεονέκτημα που έχει να προσφέρει η πολιτική μας σε αντιπαράθεση με ένα σωρά πολιτικές. Ο κύριος Πίπερ για την conditionality, τις προϋποθέσεις. Ε, βέβαια θα χρειαστούν, ε, συμφωνούμε. Τώρα για τη διαπίστευση και τις εκθέσεις ελέγχου δεν είστε ο μόνος που μου λέει ότι αυτό δημιουργεί πονοκεφάλους. Νομίζω αυτή τη βδομάδα θα γίνει μια συνάντηση με την ε, Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και τις ε, διοικητικές αρχές από τα κράτη-μέλη μας για να το ξαναδούμε με την ησυχία μας και να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Και αν μετά από τις ε, συζητήσεις αυτές και Ελπίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα λυθούν πολλά προβλήματα και από, για τις δύο πλευρές. Και τέλος θα πρέπει να συνεννοηθούμε με, βάση την κοινή λογική. Ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος. Είναι ο, αυτός που προτείνει η Κομισιόν στο δημοσιονομικό κανονισμό που θεωρείται απλοποίηση. Είναι όντως απλοποίηση. Θα επιφέρει απλοποίηση. Ή υπάρχουν κι άλλες μέθοδοι και άλλα κανάλια που θα είναι πιο αποτελεσματικά. Τώρα για τους στόχους του 2020... Όχι, αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται ακόμα. Τώρα δεν σκεφτόμαστε τόσο πολύ το earmarking, ας πούμε τη συγκεκριμένη δέσμευση κονδυλίων. Θεωρούμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ας πούμε 15-20 θεματικές προτεραιότητες που απορρέουν από τους στόχους. Και από έξυπνη, ε, διατηρήσιμη και βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Αυτά, αυτές τις ε, θεματικές θα τις παρουσιάσουμε σε εσάς. Θα συζητήσουμε μαζί σας επ' αυτών και θα αποφασίσουμε. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα σήμερα. Μετά όμως, για τα επιμέρους προγράμματα ή για τα επιμέρους κράτη-μέλη και τις περιφέρειες, ανάλογα με το, τη φύση του θέματος, θα μπορούν να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο αριθμό από τις 20 προτεραιότητες για να επικεντρώσουν τα προγράμματά τους. Στη μία περίπτωση μπορεί να είναι 2-3 προτεραιότητες που θα επιλεγούν και θα ε, προκριθούν. Σε μια άλλη περίπτωση μπορεί να είναι 5-6 προτεραιότητες. Εξαρτάται αυτό από το πόσα χρήματα θα διατίθενται. Αυτή είναι η βασική μας ιδέα σήμερα. Δηλαδή το ποιες προτεραιότητες θα επιλεγούν είναι θέμα καταρχήν των κρατών μελών και των περιφερειών. Εδώ θα ισχύει η επικουρικότητα, αλλά επικουρικότητα μέσα από διαδικασία διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην εταιρική σχέση. Πολύ γρήγορα πάω στα τελευταία θέματα που θέσατε. Σύγκληση λοιπόν σε ευρωπαϊκές περιφέρειες, κυρία Αγκουράκη, σύμφωνα με τις στατιστικές που βλέπω εγώ, μάλιστα υπάρχει κάποια, ένας βαθμός σύγκλησης, αλλά είναι πολύ βραδία διαδικασία. Θα έλεγα ψέματα να σας υποσχεθώ ότι μετά την επόμενη περίοδο θα, θα δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου όλοι θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Αλλά ο στόχος βέβαια είναι οι περιφέρειες ή μάλλον μέσα από τα αποτελέσματα να προσεγγίσουν στην ανάπτυξη και στο βαθμό ανάπτυξης οι περιφέρειες. Γι' αυτό στη μελλοντική, στην επόμενη προγραμματική περίοδο όπως και σε αυτή θα εξακολουθήσουμε να δίνουμε μεγάλη έμφαση σε ό,τι αφορά δηλαδή την κατανομή των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δίνουμε έμφαση και πάλι στις περιφέρειες εκείνες που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ανάπτυξη. Η πρόοδος όμως θα είναι βραδία. Τώρα, για τα προγράμματα που ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο όπου θα πρέπει μαζί με τις εθνικές αρχές και τις περιφερειακές αρχές να καθίσουμε και να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα να εφαρμοστούν τα προγράμματα. Γιατί μέχρι τώρα μας λέγανε ότι ναι, θα μπορούν να υλοποιηθούν. Σιγά σιγά όμως αρχίσαμε να θέτουμε σοβαρά το ερώτημα και στις περιφέρειες. Δηλαδή είναι καλό πράγμα να παραμένουν μπλοκαρισμένα λεφτά σε ένα αποθεματικό ε, για προγράμματα τα οποία ε, τελικά δεν θα εφαρμοστούν, δεν θα υλοποιηθούν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Έχουμε μερικά προγράμματα, δεν είναι πολλά, που παρουσιάζουν ε, προβλήματα αρχικά. Τώρα, για τα ε, προγράμματα ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της στέγης. Κοιτάξτε, η ενεργειακή αποδοτικότητα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι ένας τομέας στον οποίο με σχετικά μικρές επενδύσεις μπορείτε να επιτύχετε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Παράλληλα δε μπορεί αυτό να εξασφαλίσει πολύ σημαντική συμβολή σε ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς όπως την ονομάζουμε. Και βέβαια, όπως κάναμε και στα πλαίσια αυτής της προγραμματικής περίοδου και μαζί με τους συναδέλφους από το κοινωνικό μέτωπο, αλλά και από άλλους τομείς, παιδεία κλπ. Θα πρέπει να δούμε πώς θα καταπιαστούμε ε, τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων, των κοινωνικά αποκλεισμένων, με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι ακόμα και πιο μακροπρόθεσμα, ακόμα κι αν προσεγγίσουμε με πολύ έντονα εγωιστικά οικονομική σκέψη το θέμα, αλλά στο υποθέσουμε. Όταν υπάρχει μακροπρόθεσμη προοπτική θα πρέπει να δεχτούμε ότι είναι απαράδεκτο και ανυπόφορο να έχουμε 120 εκατομμύρια από τα 500 που να ζουν στο όριο της φτώχειας με φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Δημιουργείται δηλαδή εν τη αυτή περιπτώση ε, μία δυνητική αποθήκη εντάσεων που θα πρέπει να μας απασχολήσει και μακροπρόθεσμα, εξάρτητα από τα βραχυπρόθεσμα, ε, ε, από τους, μακροπρό, τους βραχυπρόθεσμους προβληματισμούς που λένε ότι κάτι τέτοιο είναι εντελώς απαράδεκτο. Σταματώ λοιπόν εδώ και ζητώ πάλι συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μπορείτε να στείλετε αυτή την περίφημη μελέτη στη γραμματεία της Επιτροπής, ε, έχει υποβληθεί. Και κάποια άλλη στιγμή μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται στις υπομετάβαση περιφέρειες, όχι τώρα, αλλά ε, ενδιαφέρει την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης το θέμα αυτό. Μα θα έχουμε συνάντηση κάθε μήνα, οπότε θα ε, μπαίνουμε και σε λεπτομερέστερα θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εξ ονόματος όλων των συναδέλφων. Τρέχουμε για να προλάβουμε το πρόγραμμα Δέκα λεπτά κυριολεκτικά έχουμε για τις εκθέσεις. Για κάθε έκθεση. Λοιπόν, δύο-τρία λεπτά η παρουσίαση και μετά να καθορίσουμε την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Δεν γίνεται αλλιώ. Πολύ γρήγορα. Η Ρόζα Εσταλά Φεραγκούτου, συγκίτρια για το πρόγραμμα στήριξη περαιτέρω ανάπτυξη μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ρόσα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εντάχει. Πρόκειται για γνωμοδότηση που αφορά πρόταση κανονισμού και ...τη διαδικασία μιας ε, ολοκληρωμένης ε, προσέγγισης για τη λήψη απόφαση και μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα που θα περιλαμβάνει το ε, βιομηχανική, περιβαλλοντική, θαλάσσια διάσταση, γιατί υπάρχουν παράκτη ζώνες που έχουν σημαντικό ελιευτικό κλάδο, επίσης άλλες που είναι σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί. Εγώ ως ε, συντάκτηρη της γνωμοδότησης πιστεύω ότι είναι σωστή αυτή η έννοια της ολοκληρωμένης πολιτικής, είναι ευπρόσδεκτη αυτή η προσέγγιση, γιατί ουσιαστικά προσπαθεί να αξιοποιήσει καλύτερα τις δυνατότητες που μας δίνει η θάλασσα. Και στη συγκεκριμένη πρόταση κανονισμού καταθέσαμε τροπολογίες που έχουν ε, τον εξής σκοπό τα, τα, τα κονδύλια που προβλέπονται που είναι 50 εκατομμύρια για τη διετή 2011-2013 θέλουμε στο μέλλον αυτή η χρηματοδότηση που είναι με πενιχρή να συνεχιστεί τουλάχιστον ώστε να εδραιωθεί αυτό το σχέδιο μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Και στις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές που θα ισχύσουν από το 2014 και μετά θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η χρηματοδότηση, περιμένοντας φυσικά χρηματοδότηση και από άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε πού θα φτάσουν τα κράτη-μέλη στην προσέγγιση αυτή, γιατί έχουν συνεργασία μεταξύ τους στον τομέα αυτό και θέλουμε φυσικά να συνεχίσουμε αυτή την, τον άξονα δράσης για να εξασφαλίσουμε και νομική ασφάλεια. Έχουμε και κάποιες τροπολογίες που προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια περιφερειακή ισορροπία για την κατανομία των διαθέσιμων κονδυλίων, ώστε να υπάρχει ένα ομοιόμορφος καταμερισμό στις διάφορες θάλασσες, γιατί άλλα χαρακτηριστικά έχει η Βόρεια Θάλασσα και άλλη Μεσόγειος. Και άλλη Μεσόγειος. Θέλουμε μια ομοιογενή κατανομή μεταξύ των κονδυλίων. Επίσης, κάποιες τροπολογίες στόχο έχουν τον έλεγχο και την επιθεώρηση, παρακολούθηση κάποιων προγραμμάτων, την εποπτεία κάποιων προγραμμάτων. Και επίσης έχουμε και κάποιες τροπολογίες για τα κονδύλια που προορίζονται για τρίτες χώρες. Γιατί με τον δημοσιονομικό περιορισμό που έχουμε χρειάζονται και τις τροπολογίες. Περιμένω και τις τροπολογίε των συναδέλφων. Δυστυχώ δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τη γνώμη και των σχεδόν εισηγητών, αγαπητοί συνάδελφοι. Οπότε τα σχόλια που θα θέλατε να υποβάλλετε σήμερα καλύτερα να τα κοινοποιήσετε άμεσα προς την εισηγήτρια. 3η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι, λίγη διορία για την κατάθεση τροπολογιών στην γνωμοδότηση της κυρίας Φεραγκούτ. Τελειώσαμε το σημείο 12 και 5 λεπτά μας απέμεινε για το σημείο 13 τη γνωμοδότηση του Λουίς Πάουλο Άλβες για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι το αντικείμενο της, δική μου γνωμο, της δικής μου γνωμοδότησης που προσπαθεί να προωθήσει τις κοινοφελείς υπηρεσίες στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας που μιλά για, τις, για τα διάφορα μέτρα, την έλλειψη νομοθετικών διατάξεων με θέμα το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Φυσικά οι κοινοφελείς υπηρεσίες έχουν κεφαλαιώδη σημασία και αποτελούν από του ακρογωνιαίου λίθους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντική η στόχη για την υλοποίηση και το, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020. Ε, συμβάλλουν στο ΑΕΠ, στην απασχόληση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και συμβάλλουν επίσης στην οικονομική ανάπτυξη και στην ενίσχυση ευημερία τη κοινωνική και εδαφική συνοχή. Οι περιφέρειές μας ε, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις κοινοφελείς υπηρεσίες και ε, γι' αυτό είναι σημαντική η συμβολή τους αυτούς και είναι σημαντικές οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης ε, θα πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η αποτελεσματικότητα στην παροχή των υπηρεσιών ώστε να επωφεληθούν οι δικαιούχοι. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικέ και να ανταλλάξουμε απόψη μεταξύ μα, αποφεύγοντας τον πειρασμό, την τυφλή και αδιαφοροποίητη εναρμόνιση μεταξύ τους. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξακριβώσει κατά πόσο τα κράτη-μέλη που προβαίνουν σε αποκέντρωση των εξουσιών προ όφελο των περιφερειακών και τοπικών αρχών για τι κοινοφιλεί υπηρεσίε συνοδεύουν αυτή την αποκέντρωση με του απαραίτητου δημοσιονομικού πόρου. Γιατί θα πρέπει ε, οι περιφέρειε να σηκώνουν το βάρο ε, ε, αυτών των κοινοφελών υπηρεσιών, ούτε να γίνουν οι περιφέρειες το θύμα των δημοσιονομικών περικοπών. Εν μέσω βαρύτατη οικονομική κρίση, σαν αυτή που διανύουμε, οι κοινοφελεί υπηρεσίε αποτελούν ένα δίκτυο προστασία για του πιο άπορους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στις ιδιωτικές υπηρεσίες. Επίσης, οι ακατοικημένες περιοχές που είναι απομακρυσμένες από τα κέντρα, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι Μαδέρια, οι Αζόρες, πολλές φορές έχουν μειωμένη ανταγωνιστικότητα και οι ιδιωτικοί φορείς δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να παρέχουν κοινοφελείς υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε αεροκατοικημένα νησιά. Σε τέτοια περίπτωση το βάρος των κοινοφελών υπηρεσιών θα πρέπει να το αναλάβουν ε, οι χώρες. Είναι πολύ σημαντική ο ρόλος αυτών των κοινοφελών υπηρεσιών. Γι' αυτό και θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερη μεταχείριση στα πλαίσια των ε, κανόνων ανταγωνισμού της ενιαίας αγοράς. Γιατί μερικές φορές δεν είναι ε, ε συνεπής η ερμηνεία που χρησιμοποιούμε χρειαζόμαστε ένα ε, σαφές επιχειρησιακό πλαίσιο και φυσικά μια νομική ασφάλεια. Μόνο με τέτοιο ισορροπημένο τρόπο θα συμφωνήσουμε με την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σεβαστεί την διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο συνεπές πλαίσιο. Περιμένω φυσικά και τις δικές σας τροπολογίες. Εγώ είμαι πρόθυμος και ανοιχτός ε, στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Λουίς. Όπω και στην προηγούμενη περίπτωση, το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλετε τα σχόλιά σα απευθεία στον κύριο Αλβε Και εδώ προθεσμία 3 Μαρτίου στι 12 το μεσημέρι. Με αυτά να κλείσω τη σημερινή συνεδρίαση ενημερώνοντα σα ότι θα συναντηθούμε σε τρει εβδομάδε. Δευτέρα 21 Μαρτίου πάλι και Τρίτη 22 Μαρτίου που και αυτή είναι πάλι πολύ φορτωμένη σε ό,τι αφορά την ημερήσια τη διάταξη. Μια γενική δήλωση. Αν θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση, αν είμαστε συντομότεροι στα σχόλιά μα, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορείτε να πείτε τέτοια πράγματα εντό δύο λεπτού, ενώ κανονικά χρειάζεται πέντε λεπτά. Και άλλοι δεν τη χάνουν τη ίδια μεταχείριση πολλέ φορέ. Γι' αυτό λοιπόν σα ζητώ να ξαναδείτε τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζετε τι συνεισφορέ σα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων μα. Ευχαριστώ πολύ και καλή σα εβδομάδα, καλή υπόλοιπο τη εβδομάδα, μάλλον.